Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας και πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα το πρωί είναι η συζήτηση για τρεις πολύ σημαντικές εκθέσεις. Η έκθεση που αφορά την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών είναι η πρώτη. Είναι η έκθεση της κυρίας Τούν und Hohenstein στη συνέχεια που έχουμε τα αποτελέσματα της εσωτερικής αγοράς και το Solvit, την έκθεση Solvit. Τρεις εκθέσεις λοιπόν. Θα δώσουμε το λόγο στους εισηγητές. Κάθε εισηγητής θα έχει τέσσερα λεπτά στη διάθεσή του για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Σας παρακαλώ να γνωρίζετε ότι στη συνέχεια οι συγητέ θα έχουν δύο λεπτά στο τέλο τη συζήτηση. Θα έχουν δύο λεπτά στη διάθεσή του για να απαντήσουν να αντιδράσουν και τρία λεπτά για την παρουσίαση. Και τρία λεπτά στην, στο τέλο, τρία και τρία έξι, διότι έχουμε και τον κανονισμό για τι δύο αυτέ παρεμβάσει. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα απ' όλα θα λάβει τον λόγο η κυρία Τούν Χόινστάιν, παρακαλώ, για να παρουσιάσει την έκθεσή τη. Έχετε τον λόγο, συνάδελφε. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, και κύριοι. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα την 19η ε, έκθεση που αφορά τις επιδόσεις ε, για την ενιαία εσωτερική αγορά και τους καταναλωτές που κατατέθηκε τον Ιούλιο περσια Αυτό το έγγραφο υπογραμμίζει και παρουσιάζει τις βελτιώσεις όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της ενιαίας αγοράς ο στόχο υιοθετήθηκε από αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι όσα ελλείμματα υπάρχουν και κατά το μέσο όρο δεν θα ξεπερνούν το 1%. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των οδηγιών που δεν υλοποιήθηκαν τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος είναι αρκετά σημαντικός. Εδώ κάνουμε λόγο για πάνω από 100 οδηγίες για την ενιαία εσωτερική αγορά και επιπλέον 22 οδηγίες δεν εφαρμόστηκαν μέσα στην περίοδο δύο ετών μετά την ε, ημερομηνία δηλαδή ε, μεταφοράς. Πρέπει να κάνουν λοιπόν περισσότερα τα κράτη-μέλη ώστε να αποτελέσει πηγή οφέλους ε, αυτή η υποβολή οδηγιών. Και σήμερα παρουσιάζω σε αυτή την οδηγία έχουμε ήδη μπροστά μας και το επόμενο scoreboard, τον πίνακα επιδόσεων, που δείχνει ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί ο μέσος όρος τώρα μη υλοποίηση είναι 0,7% ως ποσοστό το καλύτερο μέσο αποτέλεσμα ε, όσον αφορά την ιστορία μας και είναι σαφές ότι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, οι δράσεις της οδήγησαν σε μεγαλύτερη κινητοποίηση των κρατών μελών και μπορούμε να συγχαρούμε πραγματικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την συνεπή καταβολή προσπάθειας. Έχουμε και άλλα καλά μαντάτα. Όσον αφορά τον δείκτη που από το 6% πέφτει στο 5% σε αφορά την μη ε, εφαρμογή. Έχουμε κάποιες οδηγίες που δεν εφαρμόζονται σε ε, κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όσον αφορά την ύπαρξη προσκομμάτων και εμποδίων που βλάπτουν, είναι επιζήμια στην εσωτερική αγορά εις βάρος των καταναλωτών και των επιχειρηματιών. Πρέπει να καταργήσουμε αυτά τα προσκόμματα και γι' αυτό προτείνω οι φορείς και οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την ε, παρακολούθηση και εφαρμογή του νομοθετικού έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να συνεργάζονται πιο στενά μεταξύ τους. Προτείνουμε μια ε, ετήσια ε, τέτοια ε, συνάντηση ως φόρουμ θα πρέπει να διοργανώνεται. Αυτό θα δίνει την δυνατότητα στα κράτη-μέλη, στους θεσμούς, ε, στα εθνικά κοινοβούλια και στους εκπροσώπους των επιχειρηματιών και καταναλωτών να εμπλέκονται και να συμμετέχουν. Θα είναι μια καλή ευκαιρία αυτή ως βάση για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και επίσης θα συνεισφέρει να μπορέσει να δώσει στοιχεία για την κατάρτιση κατάλληλων στρατηγικών ώστε να ξεπεράσουμε αυτά τα προσχώματα. Για την άρση αυτών των προσχωμάτων ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει τα κριτήρια για την ενιαία εσωτερική αγορά εξετάζοντας πάντα τι μπορεί να γίνει σε σχέση με νέα νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζουμε ότι η νέα νομοθεσία δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις βασικές τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ενιαία εσωτερική αγορά. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι είναι για τους καταναλωτές, για τους πολίτες που δημιουργήθηκε αυτή η ενιαία εσωτερική αγορά. Και αυτή πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Επιπλέον, ζητούμε ο καταναλωτής στο πίνακας επιδόσεων της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, ο scoreboard, να δημοσιεύεται ταυτόχρονα με αυτές ε, τις ε, ε, ανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ενεπλάκησαν και προετοίμασαν, βοήθησαν στην προετοιμασία αυτής της έκθεσης και θα ήθελα να ζητήσω να υπερψηφίσετε αυτή την έκθεση. Πιστεύω ότι θα συνεισφέρει αυτή η έκθεση για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην υλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά την εσωτερική αγορά. Και σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκουν λιγότερα εμπόδια μπροστά τους και αυτό θα συνεισφέρει υπέρ τη ευρωπαϊκής οικονομίας και ταυτότητα Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και ο Πρόεδρος τώρα θα λάβει επίσης τον λόγο ως εισηγητής και για τέσσερα λεπτά η κυρία Αναχέτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους γιώδεις εισηγητές και το προσωπικό για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής μας με αυτό το θέμα. Είναι πάλι καλό το ότι έχουμε εδώ για άλλη μια φορά μια έκθεση που εκπονείται και που σίγουρα μεγάλη πλειοψηφία μπορεί να, σε μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή μας μπορεί να βασίζεται η νομοθεσία και οι προσπάθειες υπέρ των καταναλωτών πρέπει να βελτιωθούν για την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό είναι καλό τώρα το ότι από το 2007 έχουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιο για αυτό το θέμα διότι και αυτό συνεισέφερε από πλευρά του, ώστε με την πολιτική για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν να σημειωθούν πρόοδοι. Και αυτό το βαρόμετρο επιπλέον για την προστασία καταναλωτών και θέματα προστασία καταναλωτών είναι ένα αποτέλεσμα αυτή τη εργασία τη κυρία Κούνεβα. Ελπίζουμε ότι αυτό το έργο θα συνεχιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τύχει συνέχεια, ώστε τα δικαιώματα των καταναλωτών να μην αποδυναμωθούν και με τη νέα επιτροπή να ενδυναμωθούν. Είναι μια ευθύνη η οποία είναι μεγαλύτερη τώρα. Το άρθρο 12 της Συνθήκης Λισαβόνας λέγει κατηγορηματικά ότι μέσα στο πλαίσιο των διαφορετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα συμφέροντα των καταναλωτών θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη. Σημαντικό βήμα υπέρ των καταναλωτών αυτό. Και δεν θέλω να επιτραπεί τα επόμενα χρόνια να αγνοηθεί, να μεληθεί αυτή η αρχή. Χαιρετίζω λοιπόν από την άλλη πλευρά το θετικό αυτό, το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας που δημοσιεύεται με αυτόν τον τρόπο, αυτό το βαρόμετρο για την προστασία των καταναλωτών. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί πρόκειται για τα προβλήματα επίσης και τις προσδοκίες των καταναλωτών και πρόκειται για το ότι η ενιαία εσωτερική αγορά θα πρέπει να βελτιωθεί υπέρ των καταναλωτών. Η αγορά καταναλωτών στο βαρόμετρο με τους ίδιους ενδείκτες που ε, χρησιμοποιήθηκαν την τελευταία φορά εκπονήθηκε τιμή, τιμές, ε, αξιοπιστία των ε, παρόχων και ικανοποίηση των πελατών. Στο μέλλον θα εξειδικευτούν και σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθούν αυτοί οι δείκτες και νέοι δείκτες θα ενταχθούν οπωσδήποτε. Όμως όπως έχουν σήμερα τα πράγματα θεωρώ ότι αυτός ο αριθμός των δικτών είναι σωστός, ορθός και επαρκής. Διότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να κάνει και σημαντικές ε, σπουδές αναλύσεις ε, των στοιχείων. Είναι σημαντικό να δείξουμε υπομονή και να αφήσουμε χρόνο για το βαρόμετρο για να μπορέσουν να οριμάσουν τα πράγματα. Είναι ας το πω έτσι ένα παιδί που ήρθε στον κόσμο πρόσφατα και πρέπει να μπορέσει να πάρει επάνω του και να οριμάσει. Είναι σαφές επίσης ότι υπάρχουν και προβλήματα με την παροχή υπηρεσιών έναντι των προβλημάτων με αγαθά. Είδαμε ότι η διασυνορία, το διασυνοριακό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβραδύνθηκε λόγω συνοριακών προβλημάτων που οδηγούν πολλές φορές σε ανησυχία ε, τους καταναλωτές. Βλέπουμε ότι μια αποτελεσματική εφαρμογή των νομικών διατάξεων είναι, είναι σημαντικό στοιχείο και πρέπει να υπάρχει υπάρχουν δυνατότητες αποτελεσματικών ελέγχων για να μπορούν να λειτουργούν οι αγορές σωστά. Επίσης δείχνουν οι δείκτες ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και ότι υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις. Γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πράσινη βίβλο για συλλογική δυνατότητα ελέγχων, συνολικούς ελέγχους, ελέγχους να μπορέσει τη δυνατότητα να προωθηθεί. Επίσης είναι σημαντικό η ε, εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών να βελτιωθεί. Όμως οι κανονισμοί και διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ε, ομοιογενείς. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τον έλεγχο των αγορών και τους ελέγχους και τους επιθεωρητές, τις επιθεωρήσεις από πλευρά κρατών μελών. Γι' αυτό πρέπει και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν να εμπλακούν ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη και καλύτερη προστασία των καταναλωτών και να διασφαλίσουμε ότι θα αισθάνονται ασφαλείς οι καταναλωτές και θα εκμεταλλεύονται τα προτερήματα της εσωτερικής αγοράς. Είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι μηχανισμοί εποπτείας και παρακολούθησης των αγορών ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Διότι η κατανάλωση από καταναλωτών είναι εκείνο το οποίο είναι τεράστια σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κυρία Χέντ. Θα λάβει τον λόγο τρίτο συζητητή στη συνέχεια, που είναι ο κύριο Μπουσόη. Παρακαλώ. <coughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπη, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους μέχρι τώρα με βοήθησαν για να συντάξω την έκθεσή μου. Να ευχαριστήσω τα μέλη της Γραμματείας, τους κοιόδης εισηγητές και όσους ενδιαφέρθηκαν για την έκθεση αυτή και προσέφεραν στο τελικό αποτέλεσμα. Έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις που έχουν, στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη μη ορθή εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς. Είναι σημαντικό για την ίδια την αγορά, για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά προβλήματα εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων και αναζητούνται λύσεις ε, πολλές φορές ε, δικαστικές ε, στη στιγμή κατά την οποία το δικαστικό μας σύστημα είναι υπεφορτωμένο. Παρ' όλα αυτά αυξάνεται ο αριθμός των υποθέσεων που επιλύονται σε δικαστικό επίπεδο. Πάντως το τα και κέντρα αυτά τα οποία ασχολούνται με το πρόγραμμα Solvit είναι υπεφορτωμένα και αυτά με τη σειρά τους δεν έχουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν ίσως με λίγες διαφορές τα αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Αυτό βέβαια σημαίνει επιπλέον κόστος και καλούνται τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν την επάνδρωση των κέντρων Solvit και να ασχοληθούν και με εναλλακτικέ δυνατότητες χρηματοδότησης. Θέλουμε το δίκτυο αυτό να διευρυνθεί. Εγώ είμαι υπέρμαχος ενός δικτύου το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό για όλους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι μικρομεσαίες συγγνώμη, επιχειρήσεις ε, μπορούν να εξοικονομήσουν πάρα πολλά χρήματα χρησιμοποιώντας ε, την μέθοδο την οποία τους προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφεύγοντας τις δικαστικές διαδικασίες. Και φυσικά και οι καταναλωτές μπορούν να αποφύγουν διαδικασίες δικαστικές για την αποζημίωσή τους οι οποίες έχουν να απαιτούν χρόνο και χρήμα. Θα πρέπει όμως να είναι το σύστημα αποτελεσματικό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους όπως και, το και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα μέσα ενημέρωσης, τις εκστρατείες πληροφόρησης που οργανώνουν τα κράτη και επίσης να δημιουργήσουμε και μια ενιαία ιστοσελίδα Solvit. Μπορούμε να ορίσουμε κάποιον υπεύθυνο για να ασχοληθεί με την διεύρυνση του δικτύου Solvit. Σαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λοιπόν, εμείς με τη σειρά μας θα πρέπει να βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν οι συνάδελφοι στα κοινοβούλια των κρατών μελών τη σημασία αυτού του προγράμματος. Μόνο αν κατανοήσουμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το δίκτυο, τότε μόνο θα μπορέσουμε να το βελτιώσουμε και να το διευρύνουμε και να ωφελήσει ακόμα περισσότερους πολίτες. Το Solvitan ασχολείται με πάρα πολλούς συναδέλφους, με, πολλούς, με πολλές περιπτώσεις μάλλον, οι οποίες δεν εντάσσονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Και θα μπορούσαμε να προτείνουμε να υπάρξει και μία σύνδεση ανάμεσα στις ιστοσελίδες αναφορών της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αντιστοίχων επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων με την ιστοσελίδα την κεντρική αυτή του Solvit στην περίπτωση που το σύστημα δεν μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές πελάτες. Έχει τεράστιο δυναμικό το Solvit. Θα πρέπει να το αναλύουμε σωστά έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε όσο περισσότερο τις δυνατότητές του. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις των τριών εισηγητών και θα δώσουμε τον λόγο στους δύο επιτρόπους που με διαφορετικές αρμοδιότητες εμπλέκονται όμως και αφορούν τη συζήτηση που μας απασχολεί. Πρώτα απ' όλα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Μπαρνιέ. Παρακαλώ. Έχετε τον λόγο κύριε Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ε, ειλικρινά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε δίπλα με τον συνάδελφο Νταλή για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και να σας ενημερώσουμε για την εφαρμογή των διαφόρων μηχανισμών που προκύπτουν από τα νομοθετικά κείμενα. Στην πολιτική μου ζωή συχνά σκέφτομαι ότι η παρακολούθηση ενός θέματος είναι όσο σημαντική όσο η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας. Και αυτό είναι σημαντικό και στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό και στην Κομισιόν. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μέσα αξιολόγησης των πραγματικών αποτελεσμάτων των νομοθετημάτων μας για να μπορέσουμε να ενεργήσουμε σωστά στη συνέχεια και ακριβώς με αυτό ασχολήθηκαν οι συγγητές σας με πολύ προσοχή και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ ειλικρινά ε, την κυρία Τούν, τον κύριο Ζόη ευχαριστώ και την κυρία Χέρτ για την ποιότητα των εκθέσεών τους γιατί μιλάμε, γιατί πρόκειται πρόκειται για την εσωτερική αγορά αργά χθες το βράδυ έλεγα ότι σε περίοδο κρίσης στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιούμε όλα, όλες τις δυνατότητες, όλα τα ενδεχόμενα. Εάν η εσωτερική αγορά της Ευρώπης ε, λειτουργούσε σωστά όπως πρέπει να λειτουργεί, μπορούμε από μόνοι μας να κερδίσουμε ε, πρόσθετη ανάπτυξη 0,5 με 1,5% και δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή τη στιγμή αυτή την ευκαιρία. Πρέπει η εσωτερική αγορά να λειτουργεί απόλυτα σε όλες τις πτυχές της. Και ακριβώς αυτό είναι το έργο μου που μου ανέθεσε ο πρόεδρος Μπαρόζο. Γι' αυτό αποδίδω σημασία σε αυτόν τον πίνακα αποτελεσμάτων όπως και στο Solvit. Πιστεύω ότι ο Τζον Νταλή θα σας και εκείνο περίπου θα τοποθετηθεί με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τη σπουδαιότητα των καταναλωτών. Η κυρία Τούνστάιν μας εξειδίκευσε τα καλά και τα λιγότερο καλά αποτελέσματα αυτού του πίνακα αποτελεσμάτων. Υπάρχει ένα έλλειμμα στη μεταφορά σε εθνικό ε, δίκαιο. Μιλάμε για 1521 νομοθετήματα, οδηγίες, κανονισμούς κτλ. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει ένα έλλειμμα στη μεταφορά σε εθνικά δίκαιο που είναι το πιο χαμηλό από ποτέ. Αυτό είναι καλό νέο και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που στα κράτη-μέλη και καμιά φορά και στις περιφέρειες ε, έχουν αναλάβει την εφαρμογή αυτών των οδηγιών. Υπάρχει και ένα λιγότερο καλό νέο, δηλαδή η ποιότητα της μεταφοράς και της εφαρμογής δεν είναι ικανοποιητική. Συνεπώς, θα πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε, μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και τους, ε, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης ε, στα κράτη-μέλη, για να το πετύχουμε. Έχω ήδη ξεκινήσει επισκέψεις ε, προς τις 27 πρωτεύουσες, ώστε να συναντήσω τους επικεφαλείς στις δημόσιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των οδηγιών της εσωτερικής αγοράς που είναι υπεύθυνη για να λειτουργήσει το Solvit ή για τα αποτελέσματα που βρίσκονται σε αυτό το πίνακα. Συμφωνώ λοιπόν με αυτή την ιδέα ενός φόρουμ. Είναι πολύ καλή ιδέα. Πρέπει οι άνθρωποι να συνεργαστούν. Και αυτό πρέπει να γίνει ε, στο Ευρωκοινοβούλιο, με τις επιτροπές και με τους υπεύθυνους σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να ανταλλάξουμε τις καλές πρακτικές, να αξιολογήσουμε την κατάσταση και ειλικρινά πιστεύω σε αυτή την ανάγκη να συνενώσουμε τις δυνάμεις των υπευθύνων. Βεβαίως πρώτα είναι η σύμβαση και στη συνέχεια περνάμε στην κοινή εργασία. Σόλβιτ τώρα, ο κύριος Μπουζόη μας μίλησε για αυτό το μηχανισμό. 1500 υποθέσεις έχουν ε, ήδη εξεταστεί και έχουν λυθεί με διαμεσολάβευση. Πρόκειται για πολίτες αλλά και πολλές επιχειρήσεις. Ε, όλα αυτά οδηγούν σε εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Έτσι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις ε, ξαναμπαίνουν στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς αντί να περάσουν από πολύ βερούς μηχανισμούς. Ε, για να επιλύσουν τις δυσκολίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή κάποιων διατάξεων που αφορούν την εσωτερική αγορά. Μέσα στο ίδιο πνεύμα ε, έχουμε και το ΣΜΑΣ, το σχέδιο υποστήριξης για να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και στους πολίτες. Και σε αυτό το τομέα έχουν υπάρξει πρόοδοι ε, προσέγγιση μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών, ε, κοινή εξυπηρέτηση μεταξύ Solvit και ε, του μηχανισμού υποβοήθησης των καταναλωτών. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια όπως θα σας πει και ο Επίτροπος Δαλή για να παρουσιάσουμε όλες αυτές τις ανακοινώσεις, τα στοιχεία, τα αποτελέσματα ταυτόχρονα. Πράγμα το οποίο βεβαίως εξηγεί την καλύτερη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς. Συμφωνώ για αυτό το συντονισμό λοιπόν και δεσμεύομαι προσωπικά να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά όλα αυτά τα μέσα που προκύπτουν από τις 1500 οδηγίες που αφορούν την εσωτερική αγορά. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε κύριε Μπαρνιέ. Τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος που χθε είχε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε μια σημαντική, πολύ σημαντική συζήτηση για τα θέματα ισότητας και δικαιωμάτων των γυναικών. Και σήμερα με άλλο θέμα ιδιαίτερη σπουδαιότητα θα παρέμβει. Έχει τον λόγο ο Επίτροπος, παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Honorable members. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θα σχολιάσω, να μου επιτρέψετε να σχολιάσω τις δύο βασικές αυτές πολιτικές τον πίνακα αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων της αγοράς των καταναλωτών και την έκθεση heads, Να ευχαριστήσω την κυρία HEDS σαν εισηγήτρια. Η πολιτική των καταναλωτών αποτελεί τον πυρήνα των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ένας ενημερωμένος καταναλωτής, ένας ισχυρός καταναλωτής καθοδηγεί την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Ακόμα περισσότερο το να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά για τους καταναλωτές είναι το καλό μας χαρτί που θα μας συνδέσει εκ νέου με τους πολίτες. Η προσπάθεια αυτή που κάνουμε αντικατοπτρίζεται σε πολλά χαρτοφυλάκια των επιτρόπων και προσπαθούμε οι κανόνες που έχουν υιοθετηθεί να προσφέρουν πρακτικά αποτελέσματα στους καταναλωτές. Ο φίλος Μπαρνιέ, συνάδελφος Μπαρνιέ, σας έδωσε κάποιες ενδείξεις του δρόμου τον οποίο ακολουθούμε όλοι από κοινού και των πρακτικών τις οποίες χρησιμοποιούμε. Η καταναλωτική διάσταση θα πρέπει να αναπτυχθεί όπως είπα σε όλα τα χαρτοφυλάκια και να υιοθετηθούν στόχοι και επιτεύγματα για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τα βήματα πρόοδου που έχουμε κάνει. Το σύστημα αυτό ο πίνακα επιτευγμάτων είναι ουσιαστικά ένα σύστημα προειδοποίησης το οποίο μας δηλώνει τα σημεία στα οποία η εσωτερική αγορά απογοητεύει ουσιαστικά τον καταναλωτή. Πρέπει να βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά προς το συμφέρον και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του λιανικού εμπορίου γενικότερα. Πρέπει το δίκαιο του καταναλωτή να εφαρμοστεί πλήρως και να ενημερωθεί επίσης σωστά ο καταναλωτής. Για την εφαρμογή των διατάξεων χαίρομαι γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε και σε πρακτικό επίπεδο να ωφελούνται από τους νόμους, θα έλεγα και από τους διακανονισμούς και τις ρυθμίσεις που υπάρχουν γραπτά και που έχουν υιοθετηθεί στο παρελθόν. Πρέπει η εφαρμογή να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο απτή και ορατή στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω συγκεκριμένων ενεργειών. Προτεραιότητά μας είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του δικτύου το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Θα πρέπει να στείλουμε ισχυρά μηνύματα στις εμπορικές επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχουν σημαίες, ότι δεν υπάρχουν σημαίες ευκαιρίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ίδιο ισχύει και με τις αρχές των τρίτων χωρών. Για να πετύχουμε σε αυτούς τους στόχους απαιτείται τα συστήματα ελέγχου να έχουν τους πόρους και τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για να εφαρμόσουν σωστά τους στόχους τους. Σε καμία περίπτωση όμως το να προσπαθήσει να εξοικονομήσει κανείς χρήματα στα πλαίσια της μείωσης των δικαιωμάτων του καταναλωτή δεν είναι σωστό. Αυτό θα μειώσει τον ανταγωνισμό και αυτό θα είναι αρνητικό και για τον καταναλωτή και για το σύνολο της οικονομίας γενικότερα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε το μήνυμα το οποίο αποστέλουμε να το κατανοήσουν σε βάθος όλα τα κράτη-μέλη. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει στα πλαίσια των συστημάτων SWIPS, συντονισμός και έλεγχος ο συνδυασμός με τις εθνικές προσπάθειες ε, δεν είναι από μόνος του αρκετός και απαιτούνται ιδιαίτερες προσπάθειες περαιτέρω σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες που δίδει σε νομικό επίπεδο η συνθήκη έτσι ώστε να ενισχυθούν οι κοινοτικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αυτό θα γίνει εφόσον βέβαια Είμαστε πεπισμένοι ότι κάτι τέτοιο θα προσθέσει αξία στις εθνικές προσπάθειες για τα θέματα της αποζημίωσης. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα απλό σύστημα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν λάβουμε υπόψη μας τις εθνικές πραγματικότητες. Αυτό αφορά και τις συλλογικέ αποζημιώσεις. Εδώ, σε συνεργασία με τους αντιπροέδρους Σαλμούνια και Ρέντινγκ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιδείξει ικανότητα συντονισμού θα πρέπει επίσης να ζητήσω τη βοήθειά σας έτσι ώστε να έχουμε και τις απαιτούμενες πιστώσεις στη διάθεσή μας όταν εξαντληθεί χρονικά εννοώ το σημερινό ε, πρόγραμμα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και μάλιστα να βελτιώσουμε αυτόν τον πίνακα των αποτελεσμάτων, το scoreboard, και να αποδείξουμε ότι μέσα από την σωστή εταιρική μας σχέση η εσωτερική αγορά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους καταναλωτές. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τώρα θα λάβει τον λόγο για ένα λεπτό ο συνάδελφος Μπουσούτιλ που θα ομιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Έχω ετοιμάσει μια γνωμοδότηση όσον αφορά το δίκτυο Solvit και το έχουμε υποστηρίξει πλήρως γιατί είναι ένα θαυμάσιο μέσο να βοηθηθούν οι πολίτες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Θα ήθελα όμως τώρα να σας μιλήσω για την ανάγκη πλήρους συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών. Πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον πολίτη, να εξηγήσουν στον πολίτη τι μπορεί να κάνει όταν έχει δυσκολίες. Μπορεί βεβαίως να έρθει στο Κοινοβούλιο και έχουμε και το άρθρο 149 σχετικά. Επίσης, ο πολίτης μπορεί να παραπονεθεί στην Κομισιόν, στο Σόλβιτ ή και στον διαμεσολαβητή και να υποβάλει τα παραπονά του. Όλα αυτά όμως, όλα αυτά όμως περδεύουν τον πολίτη. Όταν καταγγέλει κάτι ο πολίτης δεν ξέρει πού να πάει. Εκ μέρους της Επιτροπής Αναφοράς, λοιπόν, θέλω καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών και οργάνων, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπουσούτη. Σας ευχαριστούμε που είσαστε και σύντομο στην χρήση του χρόνου στην παρέμβασή σας. Και τώρα περνάμε στους αγορητές, αγορητές που θα τοποθετηθούν εξ ονόματος των κοινοβουλευτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα η κυρία Ρόιτοβα εξ ονόματος του ΕΛΚ. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι επίτροποι, αυτή η πύλη διαδικτύου Solvit λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια και το κατάφερε 83% των παραπώνων των πολιτών ε, να τα αποφύγουμε λόγω της μη ορθής εφαρμογής των ε, όσων προβλεπόντων. Καταφέραμε μέσα σε προθεσμία 10 ημερών να διευθετηθούν αυτά τα προβλήματα. Και αυτό και κατά τη διάρκεια τη προσπάθεια αυτή, όσον αφορά τι δαπάνε ε, που, που θα προκαλούν αυτέ εξοικονομήθηκαν. Και εδώ πρόκειται για δύο προβλήματα. Πρώτον για την ελληπή εφαρμογή των όσων προβλέπονται. Πάνω από 100 οδηγίε δεν έχουν ε, ε, υλοποιηθεί ακόμα. Σημαντικό αυτό. Και το γεγονό ότι το Solvit δεν χρησιμοποιείται επαρκώ ακόμα μέχρι σήμερα. Στην Τσεχία, για παράδειγμα, μόνο 7% των επιχειρήσεων, δεδηλωμένων επιχειρήσεων γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτό το μέσο Solvit. Στην Γαλλία στην αρμόδια αρχή μόνο ένας μαθητευόμενος ε, ε, απασχολείται και πρέπει αυτό να διαδοθεί ως πρακτική το Solvit. Αυτό σημαίνει ότι τα κονδύλια από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενισχυθούν όσον αφορά το Solvit. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να γίνει πιο γνωστό το μέσο, το Solvit, να διαφημιστεί περισσότερο και να εξοικειωθούν οι πολίτες με αυτό. Είναι αναγκαίο να συνδυαστεί ε, με τις ενιαίες ε, κομβικές ε, θέσεις το Solvit να μπορέσει να συνδυαστεί με κομβικά σημεία για να λειτουργήσει καλύτερα. Είναι σημαντικό να γίνει μια ανάλυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να γνωστοποιηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Αυτή η ανάλυση θα πρέπει στην ετήσια έκθεση τη Επιτροπή να ενταχθεί ώστε να βελτιωθεί η χρήση του Solvit. Χαίρομαι για το ότι υποστηρίχθηκαν και οι τρει εκθέσει και, και πιστεύω, είμαι βέβαιο ότι θα υποστηριχθεί και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ για τη συνεργασία του ε, εισηγητέ. Ε, ε, Ευχαριστώ κυρία Ρόιτεβα. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για δύο λεπτά επίση θα λάβει τον λόγο η κυρία Γκέπχαρτ παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί κύριοι επίτροποι, Σήμερα πρόκειται για την εσωτερική αγορά, προστασία καταναλωτών, κινητικότητα των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα θέματα όταν συζητούμε για αυτά τα τρία, τις τρεις εκθέσεις και αυτά τα τρία μέσα ως εργαλεία. Και θέλω σε αυτά να επισέλθω περισσότερο. Για να συνδυάσουμε αυτά τα θέματα αν τα καταφέρουμε να τα συνδυάσουμε θα έχουμε μεγάλα ωφέλη. Πρόκειται για τα δικαιώματα των ε, πολιτών, των εργαζομένων και δεν βρίσκονται σε αντίθεση αυτά τα δικαιώματα. Πρέπει να συγκλίνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο αν θέλουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον με θετικό τρόπο. Γι' αυτό είναι καλό ότι διεξάγεται αυτή η κοινή συζήτηση σήμερα. Για να υλοποιηθούν όλα αυτά πρέπει τρεις αρχές πιστεύω, τρεις πολιτικές αρχές ιδιαίτερα να προαχθούν και να ληφθούν υπόψη. Αφενός και αυτό ο Επίτροπος Μπάρνιε πιο πριν πολύ καλά το εξέφρασε, Θέλουμε να μεριμνήσουμε ο προστατευτισμός ο οποίος είναι ιδιαίτερα ισχυρός ακόμα στα κράτη-μέλη και στις εθνικές κυβερνήσεις να ξεπεραστεί ως δεδομένο, ως κατάσταση. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτόν τον προστατευτισμό. Πρέπει να εγγραφεί αυτή η προσπάθεια στη μερίσια διάταξη. Η δεύτερη πολιτική αρχή, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι ταυτόχρονα τα δικαιώματα των καταναλωτών γυναικών και ανδρών και των εργαζομένων γυναικών και ανδρών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να διασφαλίζονται σε υψηλότατο επίπεδο. Με άλλα λόγια, η εσωτερική αγορά δεν σημαίνει κατάργηση δικαιωμάτων, δεν σημαίνει απορρίθμιση. Σημαίνει να μεριμνήσουμε ότι, ώστε αυτά τα δικαιώματα σε υψηλότερο, σε το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο να είναι σεβαστά. Και γι' αυτό κύριε και κύριοι υπάρχει ένα σημείο στην έκθεση της κυρίας Χόνσταν που δεν θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα καλό. Δηλαδή οι δείκτες ή οι επιδόσεις για την ενιαία εσωτερική αγορά. Είναι λάθος έκφραση αυτή. Δημιουργεί την εντύπωση μιας λειτουργούσας με τον τον ένα ή άλλο τρόπο εσωτερικής αγοράς πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα δικαιώματα των εργαζομένων και στα, δικαιώματα των καταναλωτών. Γι' αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή την, την έννοια όπως γίνεται στην έκθεση της κυρίας Φόνσταϊν, πρέπει να την ξεπεράσουμε αυτήν. Επίση, χρειαζόμαστε ένα πολύ καλό επίπεδο εφαρμογή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα συλλογικών προσφυγών και διευθέτηση των συλλογικών προσφυγών, ώστε οι καταναλωτέ να μην είναι μόνοι του. Ε, και να μην τους εγκαταλείπουμε, αλλά να μπορούν να βοηθηθούν. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Κυρία ε, Γκέπχαρτ, στη συνέχεια ο κύριος ε, Ρομπεροσφό. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου ξεκινώντας να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τη συζήτηση αυτή για την εσωτερική αγορά που θεωρείται μια καταπροτεραιότητα συζήτηση σήμερα. Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, κύριε Μπαρνιέ, η εσωτερική αγορά είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι ίσως ο πιο σημαντικός κινητήρας, θα έλεγα, της οικονομίας, αλλά όχι η αδίποτε μορφή κατανάλωσης. Απαιτείται μια μορφή κατανάλωσης η οποία να είναι στραμμένη στο μέλλον, να είναι αηφόρος, να σέβεται το περιβάλλον, να μην προωθεί συστηματικά τα προϊόντα discount, να μην αγνοεί την ποιότητα των προϊόντων γιατί τα προϊόντα αυτά discount είναι κακής ποιότητας και τις περισσότερες φορές είναι παρασκευασμένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θύματα πέφτουν οι καταναλωτές οι πιο εύθραυστοι με τα ασθενέστερα οικονομικά εισοδήματα. Θα πρέπει να εμπνεύσουμε μια νέα μορφή εμπιστοσύνης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στον καταναλωτή για να ενισχύσουμε και να καταστήσουμε καρποφόρα την εσωτερική μας αγορά περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Θα ήθελα να απευθύνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ντάλη, θα σας στηρίξουμε. Αλλά έχουμε όμως κάποιες ανησυχίες σχετικές με την κατανομή των αρμοδιοτήτων στα διάφορα χαρτοφυλάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας φαίνεται ότι έχει υπάρξει μια πολυδιάσπαση και διαρωτώμεθα εάν πράγματι συνεργάζεστε με σωστό τρόπο και συνεκτικό τρόπο. Θα θέλαμε τα συμφέροντα των καταναλωτών να ληφθούν υπόψη σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του πνεύματος της συνθήκης της Λισαβόνας. Ένα παράδειγμα, το οποίο δεν αφορά μόνο στους κυρίους Μπαρνιέ και Νταλή, αλλά και την κυρία Ρέντινγκ. Πρέπει να δοθεί συνέχεια στην πράσινη βίβλο για τις συλλογικέ αποζημιώσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Ντάλη αν έχετε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Θα θέλαμε επίσης να εφεύρετε μια νέα ευρωπαϊκή μορφή αυτών των συλλογικών προσπαθειών αποζημίωσης έτσι ώστε να αποφύγουμε τις υπερβολές του αμερικανικού συστήματος που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των καταναλωτών. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Χέγγ για μια πληρεστάτη έκθεση θα ήθελα να υπογραμμίσω και εγώ όπως αυτή στην εκπαίδευση για τη σωστή κατανάλωση. Αυτό πρόκειται για κάτι το οποίο δεν αφορά αποκλειστικά στους μαθητές ή τους νέους, αλλά είναι μια διαβίου προσπάθεια. Έχει, μιλάτε για τρία σχεδόν λεπτά, λέει ο πρόεδρος, άσχετο αν έχει μπλοκάρει το ρολόι πίσω μου. Να σας πω πάντως ότι ο πίνακας επιδόσεων είναι κάτι το καλό για μένα, ιδιαίτερα που είμαι στατιστικός, αλλά δεν αντικαθιστά την πολιτική βούληση που θα πρέπει να κινητοποιεί τις δυνατότητες που έχουμε. Σας ευχαριστούμε. Ήταν μια βλάβη αυτή του χρονομέτρου που απέβη προς όφελος των φιλελευθέρων. Τώρα για τέσσερα λεπτά εξ στον των Πρασίνων η κυρία Ρούλε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ίσως μπορώ εγώ να είμαι πιο σύντομη και έτσι θα αντισταθμιστεί ο χρόνος. Θα ήθελα ουσιαστικά να συνεχίσω με αυτό που είπε στην αρχή ο κύριος Μπάρνιε, τη μεγάλη σημασία της εσωτερικής αγοράς σε σημερινή κρίση. Αυτό καταδείχθηκε με σαφήνεια για άλλη μια φορά. Όμως η εσωτερική αγορά προϋποθέτει να έχουν εμπιστοσύνη φυσικά οι πολίτες σε αυτή την αγορά, στην εσωτερική αγορά. Τότε λειτουργεί αυτή σωστά. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε πολλά επίπεδα. Ακριβώς οι ευρωβουλευτές στις χώρες ε, μας βλέπουμε ότι αυτές οι φοβίες που υπάρχουν για την εσωτερική αγορά υπάρχουν ακόμα στους πολίτες μας και ότι ο προστατευτισμός εξακολουθεί να υφίσταται και δυστυχώς ε, όχι μόνο όσον αφορά τις κυβερνήσεις αλλά και όσον αφορά και τους πολίτες που υποστηρίζουν τέτοιο προστατευτισμό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό εμείς στο Κοινοβούλιο να μεριμνήσουμε να δημιουργηθεί αυτή η εσωτερική αγορά όπως πρέπει και γι' αυτό η πολιτική για τους καταναλωτές είναι κέριο στοιχείο. Κατα... Πολιτική για τους καταναλωτές, προστασία των καταναλωτών σε υψηλότατο επίπεδο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει και να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ε, χώρες μέλη την Ευρωπαϊκή Ενία Εσωτερική Αγορά. Πρέπει εδώ να καταβάλουμε ενισχυμένε προσπάθειε. Χαιρετίζω το ότι οι δύο επίτροποι ε, παρουσιάστηκαν και κατέβαλαν προσπάθειε ενωμένοι. Δεν έχουμε έναν και μόνο αρμόδιο ή μία αρμόδια επίτροπο για την ε, προστασία των καταναλωτών. Γιατί το μήνυμα που στάθηκε από την κυρία Κούνεβα ήταν πάρα πολύ θετικό και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να συνεχιστεί η προσπάθεια ε, προστασία των καταναλωτών. Να συνεργαστούμε στο μέλλον ώστε ο φόβο για την καταναλωτή κατανομή αρμοδιοτήτων σε διαφορετικούς επιτρόπους ε, και η εμπλοκή διαφορετικών επιτρόπων να ε, αποβεί ε, με θετικό όφελο και όχι εις βάρος προστασίας των καταναλωτών. Εδώ έχουμε και το θέμα για μας, το θέμα των συλλογικών προσφυγών, συλλογικών δυνατοτήτων προσφυγών. Πρέπει εδώ να μπορέσει να προχωρήσει αυτό και είναι πολύ σημαντικό για να δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη που χρειάζονται οι πολίτες. Χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα που θα καταδεικνύουν ότι οι πολίτε προστατεύονται στην εσωτερική αγορά. Ένα τέτοιο σημαντικό μέσο είναι αυτό. Και υποστηρίζουμε την ε, δυνατότητα για τις προσφυγές ε, δικαστικές ε, και αν υπάρχει δυνατότητα έξω δικαστικών ρυθμίσεων και αυτό θα ήταν θετικό. Εδώ χρειάζονται πρόσθετα μέτρα και εδώ λείπουν αυτά τα μέτρα και η εμπλοκή των, μέτρων, των μέσων αυτών στα κράτη-μέλη μπορεί να είναι μια σημαντική συμπλήρωση της, των προσπαθειών μας. Είμαι συγκίτρια για τον προϋπολογισμό μας φέτος και μπορώ να διασφαλίσω ότι τα δημοσιονομικά θέματα για την κατανομή κονδυλίων όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών θα τύχουν ιδιαίτερη προσοχή. Και από πλευρά τη Επιτροπή Προπολογισμών, τα αιτήματα που ε, λαμβάνονται υπόψη, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιούνται με το σωστό τρόπο εκεί που είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν. Μπορείτε να βασίζεστε στην υποστήριξή μα και στη συνεργασία μα. Συνολικά θέλω να πω ότι για αυτέ τι τρει εκθέσει ένα σημαντικό και πολύ καλό μήνυμα αποστέλλεται. Υποστηρίζουμε αυτέ τι εκθέσει. Ένα σημείο υπάρχει όπου πούμε επικρίσει, Τον έλεγχο για την εσωτερική αγορά, του ελέγχου. Θεωρούμε ότι είναι μονοβαρή αυτή η κατάσταση. Οι οδηγίε όταν εξετάζονται με, διαφορετικά, με διαφορετικές συνιστώσεις πρέπει να ε, εξετάζονται. Η αηφορία, τα κοινωνικά θέματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Όχι μόνο να εξετάζονται όσον αφορά την καταλληλότητά του για την εσωτερική αγορά, αλλά και για άλλε συνιστώσει ω παραμέτρους. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να υπάρχει μονοβαρή αναφορά για του ελέγχου, για την καταλληλότητα όσον αφορά την εσωτερική εσωτερική αγορά. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες ε, που γίνονται όσον αφορά την εσωτερική αγορά για να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν οι στόχοι. Και θα υπερψηφίσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Κυρία Ρούλε. Και τώρα εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών θα λάβει τον λόγο ο κύριος Μπίλαν. Δύο λεπτά παρακαλώ. Proces budowy wspólnego rynku w oparciu o cztery swobody przepływu osób, towarów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 τίματα της κοινή εσωτερικής αγοράς ώστε να πετύχουμε την υποστήριξη, την πολιτική γενικά την οποία, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ροσφόρ. Συγχαίρω τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου που ε, έδωσε προτεραιότητα σε αυτή τη συζήτηση. Και θα ήθελα να συγχαρώ και τον Μάλκολμ Χάρμπορ για τα αποτελεσματικά βήματα τα οποία πραγματοποίησε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Ε, συγχαίρω και τους τρεις εισηγητές, αλλά άκουσα και κάποια παράλογα. Συζητήσαμε την έκθεση Τούν, θαυμάσια έκθεση πρέπει να πω, για το πίνακα αποτελεσμάτων. Όμως μιλάμε για το έτος 2008. Εν τω μεταξύ η Κομισιόν έχει δημοσιεύσει τον πίνακα αποτελεσμάτων για το 2009. Είναι παράλογο αυτό. Δηλαδή μελλοντικά η Κομισιόν θα πρέπει να δίνει τους πίνακες αποτελεσμάτων ταυτόχρονα. το Solvit και τα αποτελέσματα για την προστασία των καταναλωτών ε, ασχολούνται με παρόμοια θέματα και πρέπει όλα αυτά, όλες αυτές οι ενημερώσεις και ανακοινώσει να γίνονται ταυτόχρονα. Συμφωνώ με την κυρία Τούνο ότι πρέπει να οργανώσουμε ένα ετήσιο φόρουμ για την εσωτερική αγορά και πρέπει να υπάρχουν και οι προχρεωτικές δοκιμές σε σχέση με την εσωτερική αγορά για τις μελλοντικές προτάσεις. Σας ευχαριστούμε για δυόμιση λεπτά και εξ ονόματος της Συνοπτικής Αριστεράς θα λάβει τον λόγο τώρα ο κύριος ε, συνάδελφος Φιλίδης παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει πλέον έντονη άποψη και επιβεβαιώνεται μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και από τις θέσεις της ίδιας της Κομισιόν ότι η πολιτική προστασία των καταναλωτών πρέπει να επικεντρώνεται στη διασφάλιση μιας υγιούς αγοράς μέσα από την οποία οι καταναλωτές θα δραστηριοποιούνται με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. η λογική αυτή βασίζεται στο ότι από τη στιγμή που οι καταναλωτές θα νιώθουν άνεση και εμπιστοσύνη στην αγορά και θα ενθαρρύνεται το διασυνοριακό εμπόριο θα αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα και θα δίνεται στους καταναλωτές ευρύτερη επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών σε πιο ανταγωνιστικές τιμές. η θέση και η άποψη ότι οι αποτελεσματικές και ευέλικτες καταναλωτικές αγορές αποτελούν θεμελιώδεις συντελεστές της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας των πολιτών δεν μας βρίσκει σύμφωνους. η οικονομική κρίση αποδεικνύει ότι χρειάζεται να καθοδηγούμαστε από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κράτους και όχι από δογματική μεταφορά ενός και μόνο προτύπου του ανώθευτου ανταγωνισμού. εμείς θεωρούμε ότι η ανταγωνιστικότητα δεν είναι άμεσα συνυφασμένη με την ευημερία των πολιτών γιατί πιο πολύ ευνοεί τις επιχειρήσεις αφού αποδεδειγμένα μέχρι τώρα οι των τιμών συνολικά δεν ήταν προ όφελο των καταναλωτών. θα πρέπει να υπάρξει έλεγχο των τιμών των βασικών αγαθών προ όφελο των χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων και του συνόλου των πολιτών. η μόνη πολιτική που μπορεί να θεμελιώσει και να ανεβάσει το επίπεδο προστασία των καταναλωτών είναι αυτή που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευημερία του και όχι την αύξηση του ανταγωνισμού. λέγοντα τα πιο πάνω η ύπαρξη ενός πίνακα αποτελεσμάτων που θα καταγράφει και θα αξιολογεί την ικανοποίηση των ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς μας βρίσκει σύμφωνους. από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να ξεφεύγουμε από την ουσία και τον στόχο που δεν είναι άλλος από τη λειτουργία μιας πιο ανθρωποκεντρικής εσωτερικής αγοράς στο επίκεντρο, που επίκεντρο της θα είναι η ευημερία των ανθρώπων και όχι των αριθμών αντιλαμβανόμαστε κύριε πρόεδρε την ύπαρξη ενός πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές ως ένα εργαλείο καταγραφής του δίχτυ ικανοποίησης σε συγκεκριμένο πλαίσιο και χρονικό σημείο που δεν μπορεί ωστόσο από μόνη της αυτή η αξιολόγηση και καταγραφή να επιφέρει περισσότερη ευημερία στους πολίτες απλά και μόνο επειδή κατά τα λεγόμενα θα προσδώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια στους καταναλωτές. επιπλέον η όποια αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται στη βάση κοινωνικά μετρήσιμων στόχων. σημειώνουμε επίση το γεγονό ότι αφού ο πίνακα έχει ω πρώτιστο στόχο την καταγραφή των παραπώνων των καταναλωτών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα που θα πρέπει να πάρθουν ενάντια στην αισχροκέρδεια. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε και τώρα για 1,5 λεπτό θα λάβει τον λόγο ο κύριος Ορέστε Ρώση εξ ονόματος της Ευρώπης για την Ελευθερία και Δημοκρατία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συζητάμε τρεις εκθέσεις σχετικές με την προστασία του καναλώτη. Έχουμε εκφραστεί σε σχέση με αυτό το θέμα υπέρ στις συζητήσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Επαναλαμβάνουμε τις θέσεις μας αυτές. Πάρα πολύ συχνά ο Ευρωπαίος καταναλωτής φύγεται από περιοριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναφέρομαι εδώ στην απαγόρευση ανάρτησης του Σταυρού στις ε, σχολικές τάξεις. Αυτό δημιουργεί ένα φόβο. Δεν ενημερώνεται σωστά ο καταναλωτής, ο Ευρωπαίος πολίτης για τις δυνατότητές του και τα δικαιώματά του. Θα πρέπει λοιπόν ο καθημερινός πολίτης να μην αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση τα προβλήματα τα οποία του δημιουργεί η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε επίσης και τα συστήματα ελέγχου τα οποία ισχύουν στις διάφορες χώρες. Η κυρία Τούν ασκεί κριτική στην κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα, ζητώντας να υπάρξει σωστή, κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα. Και ο κύριος Μπουσόη ζητάει να βελτιωθούν οι δυνατότητες αποκατάστασης των θυγμένων δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Τα δίκτυα τα οποία λειτουργούν σήμερα είναι ανεπαρκή και πολλές φορές οι ίδιες οι επιχειρήσεις αγνοούν την ύπαρξη αυτής της συγκεκριμένης δομής. Εμείς σαν νομοθέτες θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα λάβουμε υπόψη μας τα συμφέροντα του καταναλωτή. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Ολοκληρώνουμε αυτό το γύρο με την παρέμβαση της κυρίας Αγγέλικα Βέτμαν που θα μιλήσει για τους συναδέλφους που δεν είναι εγγεγραμμένοι. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Το Solvit μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει σημαντικά για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στην υλοποίηση και εφαρμογή όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά θα πρέπει εδώ μια πραγματιστική αρχή να ισχύει που για τους πολίτες μας αλλά και για τις επιχειρήσεις ε, χωρίς ε, μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος ε, θα διευκολύνει. Η έκθεση όμως του 2009 δείχνει ότι σχεδόν 40% των ερωτημάτων των πολιτών αφορούν διαδικασίες για διαμονή στα σε άλλα κράτη. Αυτό θέτει το ερώτημα αν υπάρχει η αναγκαία διαφάνεια ή όχι. Ευχαριστώ. Ε, Σε ευχαριστώ στον γύρο των ε, αγοριτών που ατομικά θα παρέμβουν. Πρώτα απ' όλα θα παρέμβει για δύο λεπτά ο κύριος Μότι, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Θα ψηφίσουμε την έκθεση πρωτοβουλίας για την προστασία του καταναλωτή, ένα μέσο ιδιαίτερα σημαντικό για όλους, και θα πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία Χέντ και όλους τους άλλους εισηγητές για την εξαιρετική ατμόσφαιρα στα πλαίσια της οποίας συνεργαστήκαμε. Υπήρξαν κάποια σημεία στα οποία συμφωνήσαμε πλήρως και άλλα σημεία στα οποία ελπίζω στο μέλλον να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το scoreboard, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο το οποίο όμως σε αυτή τη φάση δεν μας δίνει τα απαιτούμενα στοιχεία ομοιογένειας έτσι ώστε να μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό και να πάρουμε αποφάσεις. Αν ήμασταν μια επιχείρηση και υπολογίζαμε το τι θα κάνουμε στο μέλλον βασισμένοι σε στοιχεία τα οποία δεν είναι ενελεγμένα, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε πτώχευση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερα στοιχεία στη διάθεσή μας για να πάρουμε τις σωστές γαλήνιες αποφάσεις. Πρέπει να αυξήσουμε το βάρος του καταναλωτή, και θα πρέπει να υπάρξει και μια καλύτερη ισορροπία προς την κατεύθυνση αυτή στο μέλλον γιατί οι πολίτες δεν είναι μόνο καταναλωτές αλλά πολλές φορές είναι και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις οι οποίες συνιστούν την εσωτερική αγορά. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι δημιουργούν τις υπηρεσίες τις οποίες ο καταναλωτής αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει. Ένα σωστά ενημερωμένος καταναλωτής είναι ένας ελεύθερος καταναλωτής και από την άλλη δεν συμφωνούμε με τα εκπαιδευτικά προγράμματα γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει εμείς να υποκαταστήσουμε τον καταναλωτή και να υποκαταστήσουμε την ελευθερία επιλογής του. Ο γονιός είναι αυτός ο οποίος θα μάθει τα παιδιά να καταναλώνουν σωστά και να ελέγχουν ε, τα καταναλωτικά συνήθεια των παιδιών. Σχετικά με τους ενήλικες είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να μην είναι σωστά ενημερωμένος ο καταναλωτής. Είμαστε υπέρ των προσφυγών εξοδικαστικών όταν θίγονται τα δικαιώματά του, αλλά ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης αυτό το οποίο θα έλεγα είναι προαπαιτούμενο είναι όχι να αυξήσουμε τον αριθμό των διαμεσολαβητών, αλλά να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση σχετικά με τη δημόσια διοίκηση. Δεν έχει ληφθεί υπόψη το ότι και η δημόσια διοίκηση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο είναι πεδίο αναφοράς και προσφυγής για τον καταναλωτή. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα στο μέλλον έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που του παρέχουν τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης. Σας ευχαριστούμε κύριε Μότη για δύο λεπτά. Ο κύριος Νόκ έχει τον λόγο παρακαλώ. Merci, Monsieur le Président. Euh, euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Τούν για το, έργο της και την ποιότητα της έκθεσή της. Σαν εκπρόσωπος της ομάδας FCD S&D μάλλον, χαίρομαι που ορισμένε ιδέες ε, που θέλαμε να εμφανιστούν έχουν περιληφθεί. Τώρα, μέσα στο πλαίσιο του πίνακα αποτελεσμάτων θα θέλαμε μία προσέγγιση πιο ποιοτική ώστε να διαπιστώνονται οι λόγοι, τα αίτια της μη μεταφοράς. Ωραίοι είναι οι αριθμοί και τα στοιχεία και κάποια συμπεράσματα βγαίνουν για τους καλούς και κακούς μαθητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Κομισιόν θα έπρεπε να είναι πιο φιλόδοξη και να μετατρέψει αυτόν τον πίνακα σε μία ανάλυση των αιτίων και της δυσκολίας στην μεταφορά. Η δυσκολία στη μεταφορά. Ξέρουμε ότι καμιά φορά δεν οφείλεται στην κακή θέληση των κρατών μελών, αλλά στην κακή ποιότητα των νομοθετημάτων προς μεταφορά. Θέλουμε να ενισχύσουμε το διάλογο μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών κατά τη μεταφορά του δικαίου. Όσο περισσότερες πληροφορίες θα υπάρχουν ανάντι, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την κακή μεταφορά. Η έκθεση τώρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην παράγραφο 10. Η παράγραφος 10 δεν ήταν στο αρχικό σχέδιο της έκθεσης του. Αυτή η παράγραφος προτείνει μία δοκιμή συμβατότητας με την εσωτερική αγορά για όλες όλα τα νέα προτινόμενα νομοθετήματα. Είμαστε τελείως αντίθετοι. Ένα τέτοιο τεστ, η δοκιμή, είναι τουλάχιστον επικίνδυνο. Η εξέταση των ενδεχομένων εμποδίων για την εσωτερική αγορά πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο των μελετών που κάνει η Κομισιόν πριν ε, προτείνει νομοθετήματα. Δεν θα θέλαμε λοιπόν αυτή η δοκιμή, αυτό το τεστ για την εσωτερική αγορά να χρησιμοποιηθεί σαν πρόσχημα ώστε να παραμποδιστούν εξελίξεις για το περιβάλλον ή με κοινωνικό χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Τώρα για 1,5 λεπτό θα λάβει τον λόγο ο κύριος Κρόιτσμαν. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, το γεγονό ότι σήμερα έχουμε τρει εκθέσει ιδέα πρωτοβουλία για την προστασία καταναλωτών και για την εσωτερική αγορά και τη συζητάμε δείχνει ότι σε αυτό το επίπεδο παρόλε τι επιτυχίε πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Κατά μέσον όρο σίγουρα τα κράτη-μέλη στην υλοποίηση των οδηγιών έχουν βελτιωθεί. Παρόλα όμω, όμως αρκετά κράτη-μέλη έχουν δεν έχουν επιτύχει τον στόχο που έχει τεθεί και έτσι να μειωθεί το ποσοστό κάτω από 1% δεν είναι το κύριο πρόβλημα στην, εφαρμογή, στην εκτέλεση, αλλά στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Και έτσι έχουμε διαδικασίες για παραβίαση 18 μηνών, πολύ μεγάλη διάρκεια αυτή όσον αφορά και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο κατάσταση. Αυτές οι ελλείψεις, ε, τα ελλείμματα οδηγούν σε προβλήματα στους πολίτες και ιδιαίτερα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που εξαρτώνται από εναρμονισμένους κανόνες στην εσωτερική αγορά, όμως για κάποιους απροσδόκητους, ε, απρόβλεπτους λόγους ε, αντιμετωπίζουν προσκόμματα διασυνοριακά όταν ε, επιχειρούν διασυνοριακά. Γι' αυτό το Solvit πρέπει να επεκταθεί σημαντικά και να συνεισφέρει για την επίλυση προβλημάτων όσον αφορά και τη συνεργασία των κρατών μελών στο πλαίσιο του Solvit και έτσι με πραγματιστική προσέγγιση να επιλύονται προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή οδηγιών από τα κράτη-μέλη. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει επιτέλους να διαθέτουν αρκετά κονδύλια και κατακτισμένο προσωπικό που θα διατίθεται για τις κομβικές θέσεις Solvit. Παντού ζητάμε το Solvit στα κράτη-μέλη να γίνει πιο γνωστό, ώστε στις διασυνοριακές δυνατότητες διοχέτευσης των προϊόντων να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. Εδώ η εμπλοκή των φορέων και συλλόγων θα πρέπει να επιτευχθεί όπως και ένα ενιαίο πλαίσιο που θα μπορεί να είναι μέσα από μια πύλη διαδικτύου ένα κατανοητό εύληπτο πλαίσιο για να μπορούν οι πολίτες να το χρησιμοποιούν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ συνάδελφε. Για ένα 1,5 λεπτό τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Μάκομ Χάμπορ. Κύριε Πρόεδρε, σαν Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, με πολύ μεγάλη ικανοποίηση αντιμετωπίζουμε το ότι και οι δύο επίτροποι, οι κύριοι κύριοι Μπαρνιά και Ντάλι, είναι παρόντες σήμερα εδώ. Να υπογραμμίσω επίσης ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συζήτηση αυτή. Έχουμε μια επιτροπή η οποία κατέθεσε τρεις εκθέσεις πρωτοβουλίας που ασχολούνται με την παρακολούθηση της εφαρμογής των κοινοτικών ρυθμίσεων και όπως είπε ο Επίτροπος Μπαρνιέ τμήμα της επιτυχίας της προσπάθειας αυτής δεν θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των νομοθετικών προτάσεων αλλά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται. Αυτό είναι μια ουσιαστική εξέλιξη. Όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές θα πρέπει να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντονιστές της δικής μου επιτροπής που συνεργάστηκαν έτσι ώστε να προωθηθεί η προσπάθειά μας και να εμπλέξουμε ακόμα περισσότερο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Ελπίζω όπως ακριβώς είπατε μέχρι τώρα και οι δύο επίτροποι, ότι θα δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο φόρουμ της εσωτερικής αγοράς, να συνδυάσουμε τις εκθέσεις σας, έτσι ώστε να καταστήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα ένα ετήσιο, θα έλεγα, συμβάν σε επίπεδο επαιτειακό του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση της εσωτερικής αγοράς η οποία συγκεντρώνεται θα έλεγα σε μια πάρα πολύ συνοπτική αναφορά στη νέα συνθήκη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η πρωτοβουλία 2020 ζητάει από τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν και ακούσαμε από τους εισηγητές, τους οποίους ευχαριστώ για τις εκθέσεις του, το ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα έπρεπε να είναι μια ξεκάθαρη πρωτοβουλία και όχι να είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια μικρή παράγραφο είτε της συνθήκη είτε της πρωτοβουλίας 2020. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε συνάδελφε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό για τον κύριο Κόλμαν παρακαλώ. Τρέβορ Κόλμαν. Very much. The first note of εγώ θα είμαι η πρώτη παραφωνία σήμερα το πρωί. Αυτές οι εκτέσεις υποστηρίζουν πλήρως την εφαρμογή ε, των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και την παρακολούθηση ακόμη της ε, υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς. Ακόμη συστήνει την δημιουργία του πίνακα αποτελεσμάτων των καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια, τις καταγγελίες τους, τα παράπονά τους και μακροπρόθεσμους δείκτες. Η Κομισιόν θέλει να κάνει λοιπόν σε βάθος αναλύσεις όλων των προβληματικών αποκαλουμένων κλάδων. Αυτή η γραφειοκρατική μέθοδος ε, που θα συνεχίζει πάντοτε τις ρυθμίσεις τις κανονιστικές θα κάνουν, θα, θα καταστρέψουν τη βιομηχανία όπως συνέβη και με την Αλία παλαιότερα. Ο μικρός επιχειρηματίας πνίγεται από τις υπερρυθμίσεις της γραφειοκρατίας και όσο και χρήσιμες να είναι αυτές οι λύσεις για τους καταναλωτές, αυτή είναι ευρωπαϊκή λύση που αναζητεί προβλήματα προς λύση. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά ο κύριος Ανδρέας Σβάμπ, παρακαλώ. Με μικρόφωνο παρακαλώ κύριε Σβάμπ. Πρόεδρε, Επίτροπη, θέλω να συνεχίσω αμέσως ε, με στις σκόπιμες καλές παρεμβάσεις των συναδέλφων εκτός της τελευταίας και θα ήθελα στα πιο σημαντικά σημεία να προσέλθω. Η έκθεση της κυρίας συναδέφου Φοντούν είναι μια πολύ επιτυχημένη έκθεση ως παράδειγμα πώς μπορούμε εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο να δείξουμε ότι εννοούμε σοβαρά ότι αυτά τα οποία αποφασίζουμε από κοινού με το Συμβούλιο πρέπει να εφαρμόζονται και η εφαρμογή, η εκτέλεση είναι έργο των κρατών μελών. Εδώ πρέπει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ευρωβουλή τα επόμενα χρόνια να μεριμνήσουμε να πετύχει αυτή η εφαρμογή. Και το δεύτερο το οποίο επίσης δείχνει αυτή η έκθεση είναι το ότι ο επιμερισμός, η κατανομή όπως θέλουν να υπάρχει οι σοσιαλιστές, δηλαδή να είναι επωφελής για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει την ενιαία εσωτερική αγορά, ένας τέτοιο επιμερισμός δεν θα λειτουργήσει. Το δικό μας αίτημα είναι να ενταχθεί η εσωτερική αγορά με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα ουσιώδη στοιχεία που θεωρούν οι πολίτες ότι χρειάζονται και οι επιχειρήσεις ότι χρειάζονται να συγκλίνουν και να, να μπορούν έτσι να συλλογικά να λαμβάνουν υπόψη. Δεν θέλουμε δίσκαμπτα πλαίσια. Θέλουμε οι εργαζόμενοι να μπορούν να αγοράζουν τα προϊόντα εκείνα τα οποία εκτιμούν ιδιαίτερα. Δεν θέλουμε τις κοινωνικές δομές να τις δυσχεράνουμε στα κράτη-μέλη. Θέλουμε όμως οι κοινωνικές δομές να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο μέλλον, στις μελλοντικές προκλήσεις. Γι' αυτό πρέπει από κοινού να γίνουν οι ρυθμίσεις από την Ευρωβουλή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού. Δεν μπορεί να είναι μόνο για τι δυσκολίε αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπάρχουν μόνο ωφέλη σε σχέση με τα αιτήματα τη Ευρωβουλή. Δεύτερον, για την έκθεση αυτή που συζητήσαμε και συμπληρώθηκε από του κοιόδη εισηγητέ, δείχνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, όπως και η εμπιστοσύνη των πολιτών. Και θα πετύχει αυτό το εγχείρημα μόνο στο μέλλον, και αυτό θέλω ολοκληρώνοντα να το πω, Μόνο όταν μακροπρόθεσμα θέσουμε την εσωτερική αγορά στο επίκεντρο και αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό γενικών διευθύνσεων και τερματιστεί αυτή η αρνητική κατάσταση. Και η εσωτερική αγορά θα είναι το μεγάλο, ο μεγάλος στόχος της πολιτικής μας, κάτι που τα τελευταία χρόνια παραμελήσαμε κάπως. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι και οι δυο σας κύριοι Επίτροποι είσαστε παρόντες και αυτό θα δώσει ένα κίνητρο για τα επόμενα πέντε χρόνια που θα συνεχιστεί η προσπάθεια από την Επιτροπή στο μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Σουβάρ. Στη συνέχεια για δύο λεπτά η κυρία Στέιλερ παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αυτό και τους επιτρόπους και τους εισηγητές. Ήμουν σκιώδης για το Solvit και θα επικεντρωθώ σε αυτό το θέμα. Το Solvit είναι μια πολύ καλή έννοια και μηχανισμός. Αφορά τους πολίτες, αυτούς έχει στο επίκεντρό του και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα εμπόδια και τα προβλήματα που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λύσει τα προβλήματα μέσα σε 10 εβδομάδες. Ορισμένοι θα θεωρήσουν ότι έρχομαι από την κυβέρνηση και συνεπώς γι' αυτό το υποστηρίζω. Το Solvit όμως λειτουργεί ακριβώς υποβοηθώντας τους πολίτες. Θα ήθελα συνεπώς να τιμήσω όλους αυτούς που εργάζονται στα κέντρα Solvit, τα εθνικά. Είναι μικρές ομάδες και θα ήθελα να μιλήσω και τη μικρή ομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι υποδειγματική η λειτουργία αυτού του κέντρου. Χρησιμοποιεί το μοντέλο Solvit Plus, συν δηλαδή, και βοηθάει και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Υπηρεσία του Υπουργείου και θα ήταν πολύ σκόπιμο τα κέντρα αυτά να είναι σωστά στελεχωμένα αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Δεκέμβριο μιλήσαμε για το Solvit στην Ολομέλεια και είχα πει τότε ότι ο υπεύθυνο ε, στη χώρα σας ήταν ε, ένας νεαρός βοηθός και αυτό είναι πολύ ε, ανησυχητικό και θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι απαραίτητο τα κέντρα Solvit να είναι σωστά στελεχωμένα. Είναι σημαντικό η νομοθεσία μας να είναι σαφής και η αρμηνία της να αναπλεί για τα κράτη-μέλη ώστε η εσωτερική αγορά να λειτουργεί ομαλά και οι καταναλωτές να μπορούν να υποφεληθούν από τη βέλτιστη τιμή και υψηλή ποιότητα. Τώρα, γιατί δεν έχουμε ένα πόστερ σε, όλα μας, σε όλες μας τις περιφέρειες διαφημίζοντας το Solvit, όπως και στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ενημερώσουμε τους πολιτικούς ε, και τους τοπικούς παράγοντες για το Solvit. Ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Στήλα. Τώρα για 1,5 λεπτό θα λάβει τον λόγο ο συνάδελφος Λόκεγκόρτ, παρακαλώ. Yeah, Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι σκιώδης εισηγητής ε, για θέματα εσωτερικής αγοράς και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτό σήμερα μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας όλοι για το ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τον δίκτυ επιδόσεων για την εσωτερική αγορά. Μπορεί κανείς να δει ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα και μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα για να προαχθεί ο στόχος της εσωτερικής αγοράς, η επίτευξη αυτού του στόχου. Χαίρομαι για το ότι οι σοσιαλδημοκράτες ε, θεωρούν ότι είναι μια θετική ιδέα αυτή και ότι δεν ε, υπάρχουν, θα έλεγα, κάποιες ε, αρνητικές τοποθετήσεις. Τώρα, σε σχέση με κάποιες κοινοβουλευτικέ ομάδες που υιοθετούν κάποια διαφορετικά επιχειρήματα, μπορούμε αυτό το θέμα να το δούμε μελλοντικά. Όμως, Παρόλα αυτά, πρέπει να πω ότι χαίρομαι. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το ότι υπάρχει αυτό το συνενετικό πλαίσιο, θετικό πλαίσιο για αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να επικεντρωθώ πρώτα στο ότι καταφέραμε να καταβάλουμε τις προσπάθειες εκείνες που είναι αναγκαίες ώστε τα κράτη-μέλη στις διοικητικές τους αρχές να εμπλέκονται περισσότερο και στο εθνικό και στο περιφερειακό αλλά και στο τοπικό επίπεδο διότι αυτό που βλέπουμε να απουσιάζει είναι η αρμοδιότητα αυτών των πεδίων που πρέπει να εμπλέκονται. Υπάρχει αυτή η αρμοδιότητα και πρέπει να εμπλακούν και τότε πολλά μπορούν να γίνουν. Αναφέρθηκαν θετικά σχόλια για τα κομβικά σημεία Solvit και για την εισαγωγή μιας θέσπισης μιας ημέρας Solvit, μιας ημερίδας Solvit Καλό είναι αυτό για να εξοικειωθούν οι πολίτες που δεν γνωρίζουν το Solvit με αυτό. Και ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω. Αυτό είναι το ότι υπάρχει το γεγονός ότι πρέπει να μεριμνήσουμε εμείς και να διασφαλίσουμε και έναντι του τύπου και των δημοσιογράφων να γνωστοποιηθούν αυτά τα πράγματα, το Solvit και τον πίνακα επιδόσεων των εσωτερικών αγορών, scoreboard, για να, μπορέσει, να μπορέσουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να διαδώσουν αυτά τα στοιχεία. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια ο συνάδελφος Κοτσιούσνικ. Το πολύ. Κυρίες και πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτό που εγώ θα ήθελα να αναφέρω στην παρέμβασή μου Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρώην Επίτροπο Κούνεβα για το έργο που επετέλεσε για την προστασία των καταναλωτών και τους επιτρόπους που είναι παρόντες σήμερα, τον κύριο Μπανιέ και τον κύριο Ντάλι και που συζήτησαν μαζί μας στην Ουλευτική Επιτροπή. Να τους ευχαριστήσω για τους συναδέλφους από την Δημοκρατία της Τσεχίας που ε, συζητήσαμε μαζί. Πρέπει να πούμε ότι το Solvit είναι ένα πολύ θετικό εγχείρημα. Σε κάποιες χώρες όμως ε, η προσέγγιση του Solvit, για το Solvit πρέπει να αλλάξει κάπως και γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο ώστε οι διαφορές και όσες διαφορές υπάρχουν να ε, ξεπεραστούν και τα προσκόμματα που υπάρχουν όσον αφορά τα σύνορα να μπορέσουν και αυτά να υπερβληθούν, να τα, να τα ε, ξεπεράσουμε για να μπορέσει η εσωτερική αγορά να λειτουργήσει καλύτερα προς όφελος όλων, να υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση στην οποία βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ. κύριο παρακαλώ στη συνέχεια. Κύριε Επίτροπη, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, με την δήλωση του Επιτρόπου Μπαρνιέ στην Ακρόαση θα δώσουμε συνέχεια και θα δώσουμε ε, μεγαλύτερο, ε, μεγαλύτερη εμβέλεια στην εσωτερική αγορά. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα τότε θα πρέπει η εσωτερική αγορά να αποκτήσει ένα ενιαίο πλαίσιο. Ένα ενιαίο πλαίσιο ενιαία αγορά για να γίνει το πλαίσιο της διεξαγωγής της ζωής των πολιτών ε, της Ευρώπης. Να γίνει ο χώρος στον οποίο ζουν οι πολίτες. Να είναι ο χώρος στον οποίο ζουν ένα είδος πατρίδας. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό. Εδώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα προσκόμματα και τα εμπόδια να τα άρει και να υποβάλει προτάσεις ώστε να αρθούν. Είναι η πιο επιτυχής απάντησή μας η εσωτερική αγορά στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης προς, το εσωτερικό και προς το εξωτερικό. Η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς είναι τα προσόντα και οι ικανότητες των πολιτών μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σε τεράστιο ποσοστό συνιστούν και συναποτελούν την ε, οικονομική μας και επιχειρηματική ζωή. Γι' αυτό με το Business Act να γίνουν αυτοί οι πρωταγωνιστές της εσωτερικής αγοράς. <clears throat> Βλέπουμε ότι ε, ένα μεγάλο ποσοστό 80% ε, χρηματοδοτούνται αυτές οι προσπάθειες με πιστώσεις ε, και δάνεια και 20% με ίδια κεφάλαια. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτή τη συνιστόσα. Μετά, οι δυνατότητες εξαγωγής ε, που έχουμε και το δυναμικό μας. Πρέπει εδώ προβλήματα να τα ξεπεράσουμε και να δούμε την συνολική προσέγγιση έναντι της τομεακής, τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες έναντι των διαφορών που υπάρχουν στο κοινωνικό επίπεδο, την μονοβαρή κατάσταση ιδιαίτερα όσον αφορά το φορολογικό δίκαιο, το, τις δυνατότητες για εκπαίδευση και κατάρτιση, τις ε, δυνατότητες που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα. Χρειαζόμαστε ένα workshop για θέματα εσωτερικής αγοράς στο οποίο θα εμπλέκονται οι επιχειρήσεις ε, και με όλες αυτές τις δυνατότητες να υπάρξει μια συζήτηση αυτών των τριών εκθέσεων κάθε χρόνο, την ίδια χρονική στιγμή, την ίδια ημέρα να μπορούν να συζητηθούν ώστε η εσωτερική αγορά να γίνει το πλαίσιο ζωής, η πατρίδα των πολιτών μας. Ευχαριστώ Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κύριε Κάρας. Στη συνέχεια για ένα λεπτό η κυρία Μπερναντέτ Βερνιό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που ασχολούμεθα κατά προτεραιότητα με τις τρεις αυτές εκθέσεις που αφορούν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Συγχαίρω τους εισηγητές και θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο δίκτυο Solveit. Το δίκτυο αυτό λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια έχει επιλύσει με αποτελεσματικό τρόπο πολλά προβλήματα και παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερος παραγνωρισμένο. Πάρα πολλές φορές χρειάστηκα να παραπέμψω τους συνομιλητές μου στο δίκτυο αυτό το οποίο δεν φανταζόντουσαν ότι υπάρχει ενώ θα μπορούσε να ενισχύσει την εικόνα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών. Χαίρομαι για την παρουσία του κυρίου Μπαρνιέ. Η κυβέρνηση της χώρας μου δεν καταλαβαίνω γιατί δεν προωθεί όμως το Solvit. Η αύξηση των περιπτώσεων βέβαια προσφυγής στο Solvit θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αντικείμενο διαχείρισης για τον μοναδικό σταζιέρ που είναι υπεύθυνο για το Solvit στη Γαλλία μόνο με 60 εκατομμύρια πληθυσμό και μόνο σε δεύτερο, στη δεύτερη θέση του αριθμού των προσφυγών για τον προηγούμενο χρόνο και σχετικά με τις καθυστερήσεις 15 εβδομάδων στην αντιμετώπιση, 5 εβδομάδες περισσότερο από αυτές που προβλέπονται, είναι απαράδεκτο. Απαιτούνται χρηματοδοτικοί πόροι, απαιτούνται ανθρώπινοι πόροι, απαιτούνται εκστρατείες πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα, που το 2009 δεν υπέβαλαν περισσότερες περιπτώσεις από ότι το 2005. Σας ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό κύριος Όλε Σμιτ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη. Ευχαριστώ θερμά τους αρμόδιους εισηγητές για μια πολύ καλή δουλειά που έκαναν. Η εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη πρόοδος παρόλες τις ελλείψεις που υπάρχουν ακόμα οι επικρίσεις του κυρίου Κόλμαν δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Αυτή η πολιτική μεριμνά για καλέ θετικέ προσθέσει τιμέ και για μια προστασία των καταναλωτών που είναι καλή. Πρέπει να συνεχίσουμε σε, ε, την προσπάθεια ώστε σε ανώτατο επίπεδο να προστατεύονται οι καταναλωτέ ώστε να μπορούν να υποφεληθούν από τα ωφέλη τη εσωτερική αγορά. Αυτό είναι σημαντικό σε μια χρονική στιγμή που αυξάνεται το διασυνοριακό ε, εμπόριο και πιστεύω, είμαι πεισμένος ότι οι συλλογικέ προσφυγές θα ενισχύσουν την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Όχι όμως με το αμερικανικό πρότυπο, αλλά με το ευρωπαϊκό πρότυπο και με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι αυτό λαμβάνεται υπόψη και γίνεται αποδεκτό. Ιδίω στην παροχή υπηρεσιών εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Το γνωρίζουμε αυτό. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πετύχει την ολοκλήρωση του τομέα παροχή υπηρεσιών, ώστε να μπορεί ελεύθερα να δραστηριοποιείται η εσωτερική αγορά και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να υπάρξει γι' αυτό μια ρύθμιση για τι ε, υπηρεσίε στον τομέα υγεία με καλύτερη ποιότητα, αναβαθμισμένη ποιότητα, μικρότερο χρόνο αναμονή ε, για του πολίτε, για του καταναλωτέ. Υπάρχουν πολλέ ανασφάλειε και αβεβαιότητε και βασίζομαι σε εσά, κύριε Ντάλη, ότι θα τι ξεπεράσετε αυτέ. Υπάρχει, Πρόεδρε, υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά την, ε, ε, το θέμα των κανόνων, των διατάξεων και των κανονισμών. Όσον αφορά τι διαταραχέ τη οικονομική αγορά, γνωρίζουμε ότι αυτά δημιουργούν αβεβαιότητα και πρέπει να ρυθμιστούν. Κανόνε σαφεί είναι θετικό πράγμα για του καταναλωτέ. Σα ευχαριστώ. Ακολουθεί η παρέμβαση του κυρίου Κούρσκι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ θετικό πράγμα το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια έκθεση για το Solvit, μια έκθεση με προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Ω κοιόδης εισηγητής ε, εξ ονόματος της ομάδας ECR, πάντα είχαμε, τονίζαμε πόσο σημαντικό είναι η προαγωγή του Solvit προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ε, καταναλωτών και των επιχειρηματιών. Όλοι συμφωνούμε πιστεύω ότι το Solvit είναι μια πολύ καλή εναλλακτική μέθοδος ώστε να επιλύονται ε, προβλήματα και να διευθετούνται θέματα. Είναι πολύ θετικό, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Η εσωτερική αγορά είναι το κλειδί γι' αυτό και γι' αυτό ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υπάρξει ένας πυλώνας ε, διαδικτυακός για τα κομβικά κέντρα Solvit υπό το solvit.eu Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη την ίδια πορεία να ακολουθήσουν. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι τα εθνικά κομβικά ε, σημεία του Solvit ε, θα είναι πιο αποτελεσματικά και θα έχουν πρόσθετα στελέχη που θα εξυπηρετούν αυτά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια ο κύριος Νίτρας παρακαλώ για 1,5 λεπτό. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ όλους τους συζητητές για την προσπάθειά τους. Έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά θα έλεγα. Πρώτον, προσπαθούν να υπερασπιστούν την εσωτερική αγορά και δεύτερον, να εντοπίσουν τις αδυναμίες αυτής της εσωτερικής αγοράς. Ταυτόχρονα οι εκθέσεις αυτές είναι προτάσεις οι οποίες ε, υιοθετούνται από το σύνολο θα έλεγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακόμα και από αυτούς οι οποίοι ίσως είναι ο λίγων σκεπτικιστές σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής αγοράς. Να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω κάποια επιμέρους θέματα τώρα. Στην περίπτωση του Solvit, όπως ακριβώς είπε και ο κ. Κούρσκι, αυτό το μέσο είναι κάτι το οποίο έχει σαν στόχο να ελαφρύνει τις διαφορές που υπάρχουν ε, από χώρα σε χώρα. Αυτό ε, είναι κάτι το οποίο απαιτεί καλύτερο συντονισμό έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί πραγματικά σαν κοινό σύστημα στο σύνολο της Ένωσης. Μια άλλη σημαντική πλευρά ιδιαίτερα ε, αφορά της, την έκθεση της κόμισας Τούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να αναπτύξει ένα νέο μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η νομοθετική μας παραγωγή να μην έρχεται σε αντιπαράθεση με τις ισχύουσες συνθήκες της εσωτερικής αγοράς. Εφόσον πράγματι είμαστε βέβαιοι για την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αυτού, τότε θα είναι σε καλά χέρια η εσωτερική αγορά. Σα ευχαριστούμε συνάδελφε. Για ένα λεπτό η κυρία Μπάρμπαρα Βάιλερ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμη επιτροπή. Η υψηλή αξία που έχει η πολιτική για την εσωτερική αγορά και για τα θέματα καταναλωτών και σε αυτή την κοινή συζήτηση που καταδεικνύεται και αποδεικνύεται και η υψηλή ποιότητα και των τριών εκθέσεων. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τους συναδέλφους που επετέλεσαν αυτό το έργο. Θέλω σε δύο κέρια σημεία να επικεντρώσω την παρεμβασή μου. Το ένα από αυτά είναι το ότι εμείς ξεκινούμε από την αφετηρία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς ως Ευρωβουλή λέμε ότι όλα στην εσωτερική αγορά λειτουργούν σε ένα εναρμοσμένο πλαίσιο και έχουμε σωστές προσφορές και για τους καταναλωτές. Αυτό συχνά συμβαίνει, αλλά όχι πάντα. Υπάρχουν κάποιοι που υποβάλλουν προσφορές που είναι ανεύθυνοι και μόνο κοντοπρόθεσμα βλέπουν το κέρδος τους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ενισχυμένη εποπτεία στην αγορά και επιτήρηση Υπάρχουν όμως και μη ενημερωμένοι καταναλωτές και γι' αυτό χρειαζόμαστε καλύτερη πληροφόρηση. Δεν επαρκεί να είναι απλά αναγνώσιμα τα όσα αναφέρονται στις συσκευασίες. Χρειαζόμαστε διαρκή ροή πληροφοριών. Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη όπως αναφέρθηκε. Η εμπιστοσύνη απορρέει όμως από τη γνώση. Και στη Γερμανία άκουσα ότι μόνο κάθε δεύτερος από τους όσους είναι μεταξύ 14 και 24 ετών γνωρίζουν τι είναι πληθωρισμό, πληθωρισμός. Δεν θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη όσον αφορά το ερώτημα του αποπληθωρισμού, αν το γνωρίζουν οι πολίτες. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση λοιπόν και ε, πληροφόρηση όσον αφορά τα συμφέροντα των καταναλωτών και των πολιτών. Και αυτό σε σχέση, διακόπτει ο Πρόεδρος, ολοκληρώσατε. Και τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Στολόγιαν, παρακαλώ. Mulțumesc, domnule președinte. Este un drept Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα από τα θεμελιώτη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών είναι το εξή. Όταν θέλουν να αγοράσουν ένα προϊόν ή να εξασφαλίσουν μια υπηρεσία σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και αν βρίσκονται, πρέπει να εξασφαλίζονται αυτά από από τους ίδιους όρους, ίδια τιμή, ίδιες προμήθειες κτλ. Όταν υπάρχουν διαφορές θα πρέπει να αιτιολογούνται. Συνεπώς, νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τον χρηματοτραπεζικό τομέα, διότι αυτές τις μέρες υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην χρηματοπιστωτική αγορά στις προμήθειες των τραπεζών και των άλλων οργανισμών. Αν ζείτε, ας πούμε, στη Ρουμανία και προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια τραπεζική υπηρεσία που παρέχεται από μια τράπεζα που λειτουργεί και στη Ρουμανία και στην Ιταλία, Γαλλία κτλ. Η υπηρεσία και η προμήθεια της τράπεζας θα κοστίσει πολύ περισσότερο στη Ρουμανία και αυτό είναι πραγματικά άδικο. Πιστεύω ότι πολύ σωστά οι πολίτες αναμένουν τα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να καταπολεμήσουν αυτές τις διαφορές μεταξύ χωρών. Μιλάω λοιπόν για τραπεζικές προμήθειες, όχι επιτόκια. Ευχαριστώ κύριε Στολογιάν. Ο άλλον Κέλλη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συνάδελφους ΣΥΝΚΟΡ που ασχολήθηκαν με τον πίνακα αποτελεσμάτων. Είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολύ γιατί δίνει δυνατότητα καλής επικοινωνίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των οδηγιών. Αγαπώ αυτό το θέμα επίσης επειδή συνεχώς ακούω για υπερρυθμίσεις μέσω κοινοτικών οδηγιών στη χώρα μου, στην Ιρλανδία. Ο πίνακας αυτό σας δείχνει ότι η Ιρλανδία έχει κακοχρησιμοποιήσει τις οδηγίες σε 67 περιπτώσεις και δεν έχει, μάλλον δεν θα πετύχει και το στόχο. Ποιος φταίει όμως για αυτή της, ε, την υπερβολή στις ρυθμίσεις. Εάν δεν μεταφέρει ένα κράτος σωστά τις ε, ρυθμίσεις και τις οδηγίες, φταίει ε, η κοινότητα ή το κράτος μέλος. Νομίζω ενδεχομένως το τελευταίο. Μελλοντικά, ίσως θα πρέπει να ασχοληθούμε με την υπερρύθμιση μέσω κοινοτικών διατάξεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Τώρα έχουμε τον κύριο Σον Κέλλη για 1,5 λεπτό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ ε, αυτόν που επινόησε το τίτλο It Είναι απλός, σαφής και κάνει αυτό το οποίο λέει. Δημιουργήθηκε το 2002. Αναπτύσσεται εκθετικά, με εκθετική ταχύτητα. 22% αύξηση στις υποθέσεις εμφανίστηκε πρόσφατα και πρέπει να πω ότι οι στατιστικές είναι εντυπωσιακέ. Η άλλη πλευρά τώρα. Οι μέρες που απαιτούνται για την επίλυση ανέβηκαν από 53 σε 69 κατά μέσο όρο. Και χρειάζονται λύσεις. Ε, έλλειψη προσωπικού είπαμε. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Σωστούς πόρους, συνεχή εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη στρατηγική 2020. Ε, ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και θα πρότεινα ακόμη, επειδή πολλά από τα προβλήματα είναι τοπικά, να προσθέσουμε ένα τοπικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των καταγγελιών. Οι καταναλωτές επίσης πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα τα θέματα να ενημερωθούν δηλαδή και να έχουν περισσότερο εμπιστοσύνη. Ίσως διαδικτυακή ενημέρωση θα ήταν ε, επιβοηθητική. Τη μεταφορά τώρα των οδηγιών ε, εμφανίζονται προβλήματα και πρέπει να εξεταστούν. Συμφωνώ με τον προηγούμενο ομιλητή ότι πρέπει ε, δεν συμφωνώ μάλλον μαζί του, είναι το πρόβλημα κοινοτικό και πρέπει να βρούμε μια επιτυχημένη λύση. Σας ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό τώρα η κυρία Σιλβάνα Ράπτη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες στους εισηγητές και στους σκιώδεις εισηγητές των τριών εκθέσεων το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία με κάνει να είμαι αισιόδοξη για την πορεία της εσωτερικής αγοράς. θέλω να επισημάνω δύο σημεία. το πρώτο σημείο έχει να κάνει με την έκθεση τουν και την παράγραφο. 10. θεωρώ βασικό και νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων τα κοινωνικά δικαιώματα και η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελούν εμπόδια για την πρόοδο της εσωτερικής αγοράς. το δεύτερο σημείο αφορά το solvit. είναι ένας μηχανισμός εξαιρετικός που χρειάζεται όμως ακόμη πάρα πολύ βοήθεια και πρέπει να σας μιλήσω ειλικρινά και να σας πω ότι σκεφτόμουν να πιέσω τη δική μου κυβέρνηση στην ελλάδα να κάνει κάτι γι' αυτό γιατί διαθέτουμε μόνο δύο υπαλλήλους. όταν όμως άκουσα ότι στη γαλλία υπάρχει μόνο ένα σταζιέρ ε, σκέφτομαι να περιμένω πρώτα να πιέσει την κυβέρνησή του ο κύριος μπαρνιέ. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Και προτού περάσουμε στον γύρο των αγοριτών με τη διαδικασία Catch the Eye από πλευράς Προέδρου, θα ολοκληρώσουμε αυτό το γύρο με την παρέμβαση για ένα, 1,5 λεπτό της κυρίας ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι οι περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων λόγω κακής εφαρμογής μέσω του δεν είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα, μας δίνει αποζημίωση χωρίς τυπική διαδικασία μέσα σε λογική προθεσμία. Αυτό το δίκτυο δημιουργήθηκε το 2002, το έργο του αυξήθηκε κατά 22% το 2008. Αν και έχουμε ε, επιλύσεις 83% ε, και είναι πρέπει να σκεφτούμε να ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό δίνοντας τα μέσα να, να είναι αποτελεσματικό. Τα νέα μέτρα θα βοηθήσουν και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, ιδιαίτερα για την αναγνώριση ε, προσόντων, για κοινωνικά δικαιώματα κτλ. Το προσωπικό του Solvit πρέπει να ενισχυθεί στα κράτη-μέλη και μέτρα συνοδευτικά και εκπαιδευτικά πρέπει να ακολουθήσουν ώστε το προσωπικό αυτό να λειτουργήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είναι βασικό πιστεύω οι κυβερνήσεις και εμείς σαν ε, εκλεγμένοι των περιφερειών μας να προωθήσουμε το δίκτυο Solvit που εξοικονόμησε 32,6 εκατομμύρια ευρώ το 2008. Επίσης θα αποφύγουμε τις συνεχείς προσφυγές στο δικαστικό σύστημα. Ζητώ λοιπόν από τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν όλες τις οδηγίες και να ευαισθητοποιήσουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους με εκστρατείες ενημερωτικές. Καταλήγοντας εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας και της Επιτροπής Αναφορών, θα ήθελα η συνεργασία μεταξύ Solvit και Επιτροπής Κοινοβουλευτικής να ενισχυθεί ώστε να διευκολύνουμε το έργο όλων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκρινή. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το γύρο. Περνάμε στον γύρο των πέντε συναδέφων ακριβώς όπως προβλέπει ο κανονισμός που ζήτησαν τον λόγο στον γύρο του Catch the Eye, αυτούς που πρόσεξε και δίνει τον λόγο σε αυτούς ο πρόεδρος. Πρώτα η κυρία Χάνσλικ παρακαλώ. Ευχαριστώ τους επιτρόπους. Θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές για την εξαιρετική τους έκθεση. Προσπαθούμε να αναζωογονήσουμε την εσωτερική αγορά. Αυτό το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της ακρόασης της Επιτροπής ε, ΙΝΚΟ. Νομίζω ότι δεν έχουμε συγκεντρώσει την προσοχή μας στην εσωτερική αγορά στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εσωτερική αγορά δεν θα πρέπει να είναι κατόνομα εσωτερική. Θα πρέπει να είναι λειτουργική, καλύτερη από αυτήν την οποία έχουμε σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια σήμερα στην ελεύθερη διακίνηση θα έλεγα των υπηρεσιών και στα πλαίσια των πολιτικών προστασίας των καταναλωτών. Απαιτείται σωστή, σωστότερη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κρατημέλη. Θα πρέπει να υποστηριχθούν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας όπως το Solvit. Περνάμε στον επόμενο αγορητή. monsieur le président je ne peux que partager les conclusions du rapport de notre collègue anna id concernant. δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω τους εισηγητές σχετικά με την υποστήριξη της σωστής τάσης του καταναλωτή ιδιαίτερα σε περίπτωση όπου ο καταναλωτής είναι έφραστος οικονομικά ο πίνακα επιτυχία της κατανάλωση είναι ένα στατιστικό μέσο ενδιαφέρον μεν, αλλά ανεπαρκές, διότι ασχολείται αποκλειστικά με την κατανάλωση χωρίς να προσπαθήσει να δει ποια είναι τα προβλήματα που έχει ο καταναλωτή. Αυτός ο πίνακα δεν θα πρέπει να αρκείται στο να παρατηρεί την ζήτηση και να αφήνει τον καταναλωτή σε ένα εντελώ παθητικό ρόλο. Θα πρέπει ο καταναλωτή να παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο πιο οικολογικό ρόλο, πιο αϊφό ρόλο και θα πρέπει να υπάρξουν δείκτες και σε κοινωνικό επίπεδο και σε οικολογικό επίπεδο. Θα πρέπει να εντάξουμε επίσης στα πλαίσια της εξέτασης των νομοθεσιών. Κύριε Ευχαριστούμε κύριε, κύριε Ταραμπέλα. Στη συνέχεια ο κύριος Όντερ Μάιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφέρομαι στην προστασία καταναλωτών και τις προτάσεις που έχουν γίνει και θέλω ευθύ εξ αρχή να αναφέρω τι θετικέ πτυχέ ε, να υπάρξει αποσαφήνιση του έργου σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό, από το περιφερειακό, το εθνικό, μέχρι και το ευρωπαϊκό για τη διασυνοριακή αυτή δυνατότητα συναλλαγών και σε σχέση και με την Αυστρία. Αυτά πρέπει να γίνουν και αυστηρές κυρώσεις όσον αφορά την μη σωστή ε, κατανομή των πιστώσεων η πολιτική για τη, ε, τη σωστή κατανομή πιστώσεων είναι σημαντικό. Επίσης εδώ όσον αφορά το δίκαιο και την ε, δυνατότητα προσφυγών που σε εμά στην Αυστρία μέσα σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο ε, εντάσσονται και να δούμε και τις ε, εθνικές ρυθμίσεις που μπορούν να προστατεύουν καλύτερα τους καταναλωτές. Θα πρέπει όταν υπάρχει ανάγκη αυτά να χρησιμοποιούνται ως μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια κυρία Μαγκίνες. Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προστασία των καταναλωτών ευνοείται από όλους μας. Το πρόβλημα είναι ότι λόγια-λόγια από ορισμένα κράτη χωρίς να γίνονται πολλά πράγματα για το Solvit. Δεν έχει προσωπικό. Θα σας δώσω ορισμένα προβλήματα το που αντιμετωπίζω στο γραφείο μου. Ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι η μεταβίβαση δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν και τους αλλοδαπούς όπως τους ιδιούς πολίτες τους. Χρειάζεται κάτι να γίνεται. Ε, ε οδηγοί επιχειρηματικοί, τα city guides ας πούμε, ε, εξακολουθούν να μου δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν, διότι η στάση των πολιτών σε σχέση με την εσωτερική αγορά επηρεάζεται από τις εμπειρίες τους, ακόμη και αν δεν είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε με την παρέμβαση της κυρίας Σαρλεμόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συζήτηση που έγινε εδώ σήμερα. Χαίρομαι για το ότι ο κύριος Μπαρνέ και ο κύριος Νταλή οι επίτροποι υπεγράμμισαν από πλευρά του ότι χρειάζεται υποστήριξη από πλευρά μα για την επίτευξη τη εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ιδιαίτερο ειδικό σημείο στην έκθεση τη κυρία Head, το σημείο 40. Εκεί σε αυτό προτείνεται μια ευρωπαϊκή υπηρεσία για τους καταναλωτές να δημιουργηθεί. Θα ήθελα να ακούσω επ' αυτού αν οι επίτροποι θα δώσουν συνέχεια σε αυτό το αίτημα διότι θα μπορούσαν μελέτες να συνταχθούν για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, για παράδειγμα. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει βάση για το έργο, ε, την εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου σε σχέση με θέματα καταναλωτών. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας, Επίτροπη. Θα δώσετε συνέχεια σε αυτό ως θέμα, διότι θα μπορούσα να φανταστώ ότι μια τέτοια υπηρεσία θα μπορούσε να έχει την έδρα της είτε στη Μάλτα είτε στη Γαλλία. Πρόεδρος, ολοκληρώθηκε ο γύρος των παρεμβάσεων και όσον αφορά τη διαδικασία κάτω DI από πλευρά Προέδρου και τώρα θα δώσουμε τον λόγο στου δύο επιτρόπους για να τοποθετηθούν στι διαφορετικέ παρεμβάσει των Ευρωβουλευτών που έγιναν. Πρώτα απ' όλα θα λάβει τον λόγο ο επίτροπο κ. Μπαρνιέ, παρακαλώ. Ε. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Η κυρία Σαλντεμόζε υπογράμμισε την ποιότητα που χαρακτήρισε τη συζήτησή μας και να πω ότι η υπηρεσία των καταναλωτών υπάρχει και θα πρέπει να σχολιαστεί καλύτερα και από μένα και από τον κύριο Ντάλη. Συμφωνώ πάντως με την αξιολόγηση που έγινε για την ποιότητα της συζήτηση που προηγήθηκε για τις επικοδομητικές προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά με την αξιολόγηση και την ε, παρακολούθηση αυτών των 1500 οδηγιών και διακανονιστικών κειμένων, επαναλαμβάνω τον αριθμό 1500 που οργανώνουν και χαρακτηρίζουν την εσωτερική αγορά. Και προτιμώ να μιλάω για μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά και όχι για ενιαία αγορά. Αυτό θα το καταλάβει καλύτερα ο καταναλωτής πολίτης. Ελέγχομαι εδώ από τον κύριο Χάρμπορ γιατί το είπα αυτό και στην επιτροπή του. Όπως επίσης και στην παρέμβαση του κυρίου Τριαφελίδη. Να υπενθυμίσω ποια είναι η πορεία την οποία θα ακολουθήσω εγώ και η Επιτροπή τα επόμενα πέντε χρόνια. Πρόθεσή μου, κυρίες και κύριοι, μέρα με τη μέρα και νομοθετική ρύθμιση μετά από νομοθετική ρύθμιση είναι η εσωτερική αγορά να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών ανδρών και γυναικών που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη φιλοδοξία είναι μια και είμαι υπεύθυνο για τις αγορές ή χρηματαγορές για τις οποίες μιλάμε πολύ τους τελευταίους μήνες να υπηρετούν την πραγματική οικονομία, τους πολίτες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει οι καταναλωτές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να ξαναμπούν σε αυτή την αγορά. Αυτές είναι οι δύο κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες θα ακολουθήσω στα πλαίσια του συνόλου των επιτρόπων. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και επανέρχομαι εδώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ροσφόρ και άλλοι προηγουμένως. Είναι θέμα αμοιβαία εμπιστοσύνης και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία ε, Φοντούνου Χέρχενστάιν για την ποιότητα της εκθέσεώς της σχετικά με τον πίνακα επιτευγμάτων ή αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς. Στην έκθεση αυτή υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω. και άλλοι υπογράμμισαν την μεγάλη σημασία των δικτών τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια της εκθέσεως Φοντούν. Η κυρία Γκέμπχαρτ αναφέρθηκε στην κοινωνική διάσταση και στην οικονομική διάσταση των οδηγιών. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα λίγο να ανταποκριθώ και στην επικοδομητική κριτική του Μάλκομ Χάρμπορ σχετικά με τη στρατηγική γύρω από το 2020. Και η κυρία Χάντσλεκ είπε ότι δεν μιλάμε πολύ για την εσωτερική αγορά. Αν διαβάσετε προσεκτικά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, η εσωτερική αγορά είναι παντού έξυπνη ανάπτυξη, ευρεσιτεχνίες, άλλα μέσα, πράσινη ανάπτυξη με τη σωστή χρήση των δημοσίων προμηθειών, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη ανάπτυξη, παντού βρίσκεται η εσωτερική αγορά, οφείλει να βρίσκεται παντού η εσωτερική αγορά. Και βέβαια να μην ξεχνάμε όμως ότι η έκθεση 2020 δεν αναφέρεται στα πάντα, δεν αναφέρεται στην άμυνα, δεν αναφέρεται στην εξωτερική επιτροπή και δεν θα υποκαταστήσει την εργασία την οποία επιτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι θεματοφύλακας και παρακολουθεί σωστά το, την εφαρμογή των κειμένων των δεσμευτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένας από τους στόχους μου και πολλές φορές θα χρησιμοποιώ και τις διαδικασίες επί παραβάση έτσι ώστε να εφαρμοστούν σωστά οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Πάντα όμως θα προκρίνω την εμπιστοσύνη, τη συνομιλία, το διάλογο και όχι τόσο τον εξαναγκασμό. Στην έκθεση της κυρίας Χόχενστάιν Φοντούν υπάρχουν και άλλες πολύ καλές ιδέες όπως η συνεργασία με τα κράτη-μέλη και η δημιουργία του Φόρουμ της Εσωτερικής Αγοράς το οποίο υποστηρίζω. Και, ως, και μάλιστα τη στιγμή που θα δημιουργηθεί ίσως να το συνδυάσουμε και με άλλες πρωτοβουλίες στα πλαίσια του ίδιου θέματος που συζητάμε με τον Τζον Ντάλι, τον άλλο επίτροπο. Παράδειγμα, η αξιοστότερη αξιοποίηση του δικτύου Solvit. Δίνω πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο στην ανακοίνωση ενός προγράμματος αλλά και σωστή εφαρμογή του και παρακολούθησή του. Γι' αυτό αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων θα μας επιτρέψει όχι μόνο σε ποσοτικό επίπεδο να παρακολουθήσουμε το πόσες οδηγίες εφαρμόζονται, αλλά και σε ποιοτικό επίπεδο. Ο κύριος Χουάνγκ Νοκ είπε πάρα πολύ σωστά ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η ποιότητα της εφαρμογής και της μεταφοράς των κοινοτικών νομοθετημάτων σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό φυσικά για ένα επίτροπο θα έλεγα είναι μια πάρα πολύ σωστή άσκηση θα έλεγα ελέγχου. Αυτά. Ευχαριστώ όλους που υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες αυτές όπως ο κύριος Σουάμπ και η κυρία Ρόικα. Για το Solvit τελειώνοντας με κάποιες πρώτες εκτιμήσεις συνοπτικότατες. Συμφωνώ με αυτούς που είπαν ότι απαιτείται να υπάρξει μια ιστοσελίδα solvit.eu. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μια ιστοσελίδα που θα παραπέμπει στις εθνικές ιστοσελίδες. Επεξεργαζόμαστε αυτή την πρόταση πάρα πολύ ε, ε, ενεργά. Και όπως είπε και ο Σον Κέλλη, Mm. Έστω και η λέξη it λέει τα πάντα. Είναι πάρα πολύ απλή και ξεκάθαρη η λέξη. Και νομίζω είναι μια πρώτη θετική κριτική. Το it δουλεύει, δουλεύει καλά, θα μπορούσε να δουλεύει καλύτερα όμως. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες και πάρα πολλές επιχειρήσεις που αγνοούν τα δικαιώματά τους και τον τρόπο προστασίας αυτών. Και εδώ έρχομαι σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Βέρκμαν η οποία ζητά να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια. Νομίζω ότι πολλοί από εσά, κυρία Βερνιό, κύριο Γρόση, Στήλερ, Ράπτη, αναφέρθηκαν στην ανεπάρκεια των μέσων που έχει στη διάθεσή του το σύστημα Solvit. Και όχι μόνο στη Γαλλία βέβαια, αν και άκουσα πάρα πολύ καλά αυτά που είπατε για τη Γαλλία. Και εγώ δεν ομιλώ εδώ σαν υπουργό, αν και ήμουν παλαιό υπουργό. Και δυστυχώ γνωρίζω πολύ καλά τι συμβαίνει στη χώρα μου, πάντα χώρα μου είναι, και τι δεν πάει καλά. Πράγματι απαιτούνται περισσότερα μέσα και θα τα ελέγξω όλα αυτά στα πλαίσια των επισκέψεων τις οποίες θα κάνω επί τόπου. Λοιπόν, τα μέσα αυτά όπως είπαμε είναι απαραίτητα για να δούμε πώς δουλεύει η εσωτερική αγορά. Αυτή η εσωτερική αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να αναζωογονηθεί να εμβαθυθεί, το είπανε πάρα πολύ καλά ο κύριος Κάρας, η κυρία Γκέπχαρτ, ο κύριος Σόλου Σμιτ και σε επίπεδο διαμεθοριακό και σε επίπεδο εσωτερικό κάθε χώρας πρέπει να αρθούν τα εμπόδια που υπάρχουν. Ίσως αυτό να μην υπογραμμίζεται επαρκώς, αλλά συμπεριλαμβάνεται στη στρατηγική του 2020 να βρούμε πού υπάρχουν τροποπέδες και να τις απομακρύνουμε και θα συνεργαστώ με τους 12 συναδόλφους επιτρόπους οι οποίοι ασχολούνται και αυτοί με τον ένα τρόπο ή τον άλλο με την εφαρμογή των οδηγιών στην εσωτερική αγορά. Τρεις συγκεκριμένες παρατηρήσεις τώρα. Ναι, όπως είπε ο κύριος Μπούσετιλ, ναι σε μια στενή συνεργασία ανάμεσα στον Ombudsman, στο Solvit και στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Ρούλε και όλους τους άλλους από την Επιτροπή Προϋπολογισμών για την ε, θέλησή τους να υποστηρίξουν το Solvit δημοσιονομικά. Ευχαριστώ επίσης και την κυρία Γκρούνη για τα σεμινάρια τα οποία ζήτησε να δημιουργηθούν ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους στα διάφορα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες μερικές φορές που ασχολούνται με το Solvit. Και τέλος, ένα θέμα το οποίο έγινε αντικείμενο κριτικής από τη σοσιαλιστική ομάδα. Θα πρέπει να αποδραματοποιήσουμε το θέμα αυτό του ελέγχου της εσωτερικής αγοράς. Κάθε νομοθετική πρόταση που περνάει και από εσά θα πρέπει να σέβεται τη συνθήκη. Αυτό θέλει να πει η συγγήτρια. Θα πρέπει να περνάει ένα τεστ ελέγχου συμβατότητας με τις βασικές εδρεωμένες αρχές της εσωτερικής αγοράς θα προσπαθήσω έτσι ώστε από εδώ και πέρα κάθε νομοθετική ρύθμιση να αξιολογείται εκ των προτέρων σε σχέση με ορισμένα κριτήρια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά. Αυτή είναι η ανάληψη υποχρέωση την οποία δηλώνω, έτσι ώστε και από πριν και εκ των υστέρων θα πρέπει όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις να γίνονται τμήμα του νομοθετικού κόρπους που εξυπηρετεί τον πολίτη και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο έδαφος της Ένωσης. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε Μπαρνιέ. Τώρα ο Επίτροπος Νταλή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως και ο συνάδελφός μου, Μισελ Μπαχνιέ, είναι πολύ χρήσιμο να είναι κανείς σε μια, παρόν σε μια τέτοια συζήτηση τόσο ε, ενδιαφέρουσα που έχει σχέση με τους καταναλωτές. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε όλοι με πραγματικό πνεύμα συνεργασίας ε, και να βάλουμε σαν πρώτο στόχο τους την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Επανέρχομαι σε κάτι που είπα στην εισήγησή μου. Εκτός από τα οικονομικά επιχειρήματα για μια σωστά εφαρμοσμένη και αποτελεσματική πολιτική για τους καταναλωτές, δεν πρέπει να ξεχνάμε το κεντρικό σημαντικό ρόλο που μπορούμε να παίξουμε για την επανασύνδεση της Ευρώπης με όλους τους πολίτες της. Είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο αυτό. Ξέρω ότι πρέπει να συντονίσω αυτό το έργο είναι μέσα στα καθήκοντά μου και η επαγρύπνησή σας θα με συνοδεύει, το γνωρίζω. Ο πίνακος αποτελεσμάτων μας δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε αποτυχίες στην αγορά, και μας δίνει ακόμη τη δυνατότητα να τις αντιμετωπίσουμε αυτές τις αποτυχίες. Είναι κρίσιμος αυτός ο μηχανισμός. Έχει πραγματικά στόχο και μπορούμε να ωφεληθούμε από την περαιτέρω ενίσχυσή του. Ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι τα μάτια μας και τα αυτιά μας που μας ξυπνούν στα προβλήματα και είναι κοινή η δέσμευσή μας για αποτελεσματική εφαρμογή των ρυθμίσεων ώστε να ενισχύσουμε τον Ευρωπαίο καταναλωτή και να υπάρξουν τα σωστά οικονομικά ωφέλη. Μετά από μια δημόσια διαβούλευση πέρυσι η Κομισιόν αξιολογεί τα σχόλια σε σχέση με τις συλλογικές αποζημιώσεις και προτίθεται να βρει λύση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών χωρίς να φτάσουμε σε αμερικανικές λύσεις. Η εναλλακτική επίλυση των διαφορών είναι η κινητήρια δύναμή μας. Ο συνάδελφος και φίλος Μπαρνιέ ε, εξήγησε τη στρατηγική 2020 για την εσωτερική αγορά. Αν κοιτάξετε από κοντά τα κείμενα θα δείτε ότι οι καταναλωτές πρέπει να μείνουν στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς. Είναι η κινητήρια δύναμη της ενιαίας αγοράς και πρέπει να ενισχύσουμε την κεντρική τοποθέτηση των καταναλωτών. Όσον αφορά την παιδεία των καταναλωτών, πράγματι είναι ένα θέμα κλειδί αυτό και πρέπει να δούμε πώς το πρόγραμμα Dolcetta μπορεί περαιτέρω να ενισχυθεί, να καλύψει νέους τομείς. Όσον αφορά το τελευταίο σχόλιο σας για τον οργανισμό για τους καταναλωτές, η εφαρμογή των διατάξεων είναι υποχρέωση του κάθε κράτους και πρέπει το κράτος να παρέχει τους απαραίτητους πόρους. Όμως υπάρχει και νομική βάση για τη συμπλήρωση των κονδυλίων ε, από την πλευρά της Ένωσης. Και πρέπει συνεπώς να αναζητήσουμε τις βέλτιστες λύσεις, τις θεσμικές και τις οργανωτικές και η Κομισιόν θα εξετάσει όλες τις εναλλακτικές προτάσεις. Ε, ελπίζω ότι θα κάνουμε μεγάλη πρόοδο όσο χρόνο θα μείνω υπεύθυνο για αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντάλι. Κυρία Τούν Χόχενστάιν για τα συμπεράσματά της. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για τις παρατηρήσεις σας. Ακούσαμε τις απόψεις και των δύο επιτρόπων. Βλέπουμε λοιπόν ότι το νέο Κοινοβούλιο και η νέα Επιτροπή θα μπορέσουν να συνεργαστούν αποτελεσματικά και στενά για να αναπτύξουν περαιτέρω την εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά, η ενιαία αγορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις θετικές αντιδράσεις στις προτάσεις μου στην που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Οι συνάδελφοι της Σοσιαλιστικής Ομάδας ανησυχούν για την παραγράφο 10 και για τη δοκιμή ενιαίας αγοράς. Σας με θυμίζω ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Αυτή η πρόταση ε, εγκρίθηκε το 2003 από την Επιτροπή ΙΝΚΟ είναι μέρος της στρατηγικής της εσωτερικής αγοράς. Μην ανησυχούμε, δεν πρόκειται να καταργήσει την κοινωνική πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος μόλις αναφέρθηκε στο γεγονό ότι κάθε νέο νομοθέτημα αξιολογείται σε σχέση με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος για πανικό. Όλοι θέλουμε την εσωτερική αγορά να ενισχυθεί, να εξελιχθεί ε, ε, Θέλουμε να μείνουμε μακριά από τις ε, τάσεις προστατευσισμού. Η ολοκλήρωση της Ευρώπης μπορεί να υλοποιηθεί μόνο όταν οι πολίτες έχουν συνείδηση των πραγμάτων και η δημόσια διοίκηση είναι φιλική προς τους πολίτες. Η έκθεση μου λοιπόν προτείνει διάφορες λύσεις. Λύσεις που θα βοηθήσουν τους εκλογείς μας να συμμετάσχουν περισσότερο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ε, η εσωτερική αγορά είναι το μεγάλο επίτευγμα, επαναλαμβάνω. Πρέπει συνεπώς να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς που θα υποστηρίξουν αυτή την ενιαία αγορά. Η δημοσίευση των τεσσάρων εκθέσεων είναι βεβαίω σημαντικό στοιχείο και ένα βήμα προς τα πρόλη Ας μην γινόμαστε αλλεργικοί προς την έννοια της αγοράς. Ε, από το χώρο από τον οποίο εγώ προέρχομαι είχαμε, περάσαμε πολλές δεκαετίες κατά τις οποίες δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε καθόλου για ελεύθερη αγορά. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα τώρα όμως. Οι ελευθερίες είναι στην καρδιά της ενιαίας και κοινή μας αγοράς. Και ας εξασφαλίσουμε να μην περιορίζονται αυτές οι ελευθερίες. Ας βοηθήσουμε τους πολίτες μας να ενισχυθούν από αυτές τις εξελίξεις. Η κυρία Χέντ τώρα, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς όλες τις ενδιαφέρουσες ε, παρατηρήσεις και συνεισφορές. Χαίρομαι που οι δύο επίτροποι ε, υποσχεθήκαν ότι θα συνεργαστούν για να ενισχύσουν την προστασία των πολιτών περαιτέρω. Οι οργανώσεις των καταναλωτών έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν, πρέπει να σας πω. Όταν ειδικότερα πρόκειται να προσελκυθεί η προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε σε αυτές τις οργανώσεις καταναλωτών για να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά εθνικά. Ακόμη, τα κράτη-μέλη πρέπει να παροτρινθούν να επιζητήσουν τη συμμετοχή των, οργανισμών, ε, των οργανώσεων καταναλωτών για τα θέματα που αφορούν τους καταναλωτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Νταλή ε, που ε, τόνισε ότι θα, προχωρεί, θα προσπαθήσει να επιτύχει τη σωστή επάντρωση αυτών των κέντρων για να ενισχυθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων. Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι ο ε, πίνακας αποτελεσμάτων πρέπει να βελτιωθεί όχι μόνο σε σχέση με την πολιτική για τους καταναλωτές, αλλά πρέπει να επιδράσει σε όλες τις πολιτικές που επηρεάζουν τους καταναλωτές. Άρα θα πρέπει να εντάξουμε την πολιτική για τους καταναλωτές σε όλο το φάσμα των κοινοτικών πολιτικών ώστε αυτά τα θέματα να ρυθμίζονται και στο κοινοτικό και στο εθνικό επίπεδο. Ε, θα επανέλθουμε σε ένα χρόνο ελπίζω σε αυτό το θέμα και θα το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούσο, η τελευταία συζήτηση, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μπαρνιέ και τους συναδέλφους που ε, επένεσαν την έκθεσή μου και μίλησαν θετικά για το δίκτυο Solvit. Είναι πρακτική λύση για τους καταναλωτές το δίκτυο Solvit και γι' αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και να τον ενισχύσουμε και να το καταστήσουμε γνωστό σε όλους τους καταναλωτές. Έτσι οι καταναλωτές θα μπορέσουν να προασπίσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους. Τα αποτελέσματα που πετύχαμε στην Επιτροπή Αναφορών και Εσωτερικής Αγοράς είναι ικανοποιητικά. Το Solvit λειτουργεί ήδη σαν δίκτυο, αλλά θα πρέπει να επιλύσουμε κάπως τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν αυτοί που χρησιμοποιούν το Solvit και το, ε, τα στελέχη που το επανδρώνουν. Αναφέρθηκαν πολλές λύσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την καλύτερη επάνδρωση. Βεβαίως χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό σε αυτά τα κέντρα και το προσωπικό αυτό θα πρέπει να έχει τα σωστά προσόντα, να έχει την κατάλληλη κατάρτιση για τους κανονισμούς και τις οδηγίες και τις ρυθμίσεις. Πρέπει επίσης το προσωπικό αυτό να τύχει της νομικής στήριξης της δημόσιας ε, και της Κομισιόν, επειδή πρόκειται για περίπλοκες περιπτώσεις. Η, ε, καμιά φορά η Κομισιόν παίρνει πολύ χρόνο για να απαντήσει στα αιτήματα της Solvit. Θα ήθελα να επιταχυνθεί αυτό και ευχαριστώ τον ε, Επίτροπο Μπαρνιέ που είπε ότι το ταχύτερο δυνατόν θα ανεβάσει τη διαδικασία την δικτυακή πύλη για το Solvit. Πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει την καλή λειτουργία του δικτύου και καλώ όλες τις ομάδες να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουσουτσόη. Πέρας λοιπόν της ε, συζήτησης, η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στις 12. Ευχαριστούμε και εσάς και τους επιτρόπους. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του Κάρλος Κοέγιο σχετικά με την κυκλοφορία προσώπων με θεώρηση μακράς διαμονής.